Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, καλεσμένοι, καλεσμένοι μας. Ε, σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρία της Επιτροπής Γυναικών. Δυστυχώς ακολύεται σήμερα η Πρόεδρος, οπότε θα προεδρεύσω εγώ. Σήμερα είναι μήνυμα από τις Διερμηνείς. Βρισκόμαστε στην 35η μέρα των, δια, των διαμαρτυριών μας κατά της μονομερούς επιβολής από τη Διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άδικων συνθήκων εργασία στου διερμηνεί. Με τα λύπη σα πληροφορούμε ότι η διερμηνία θα διακοπεί στι 6.30 ακριβώ, δηλαδή την προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη, λέει ο πρόεδρο. Ε, υπάρχουν προτάσει για αλλαγέ. να θεωρήσω ότι εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Okay, the second point is... Uh, Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Δύο συνεδριάσεων. Αν δεν υποβληθούν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ξεκινάμε με τις συστάσεις των συντονιστών. Στη συνεδρίαση της 20ης ε, Ιουνίου, οι συντονιστές αποφάσισαν τα Να καταρτήσουν έκθεση με τη μορφή τροπολογιών στην ομοθετική έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τα στατιστικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και να την αναθέσουν στην ομάδα φιλελευθέρων. Επίσης, θα εκπονήσουν γνωμοδότηση στην ε, μη νομοθετική έκθεση τη Επιτροπή Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική σχετικά. Την ανέλαβε το ΕΛΚ. Επίση, ε, σύνταξη γνωμοδότηση στη μη νομοθετική έκθεση τη Επιτροπή Απασχόληση για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο ανατέθηκε στου Πρασίνου και επίση ε, με τη μορφή τροπολογιών θα συντάξουμε τη θέση μα ε, και θα την επιδώσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ που είναι αρμόδια καθήλη για την έκθεση με το ίδιο θέμα. Την ανέλαβαν οι σοσιαλιστές αυτή τη σύνταξη των τροπολογιών. Επίσης δεν υπάρχει αποχρόν λόγος για να συμβάλλουμε ως Επιτροπή Γυναικών στην Ομοθετική έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση των τεχνολογιών για την υγεία. Επίσης, θα συντάξουμε προφορική ερώτηση με ψήφισμα για τις, πολιτι... για τις προκλήσεις και τις στρατηγικές ε, ε, σε ό,τι αφορά τους γυναικείους καρκίνους και τις συναφείς νοσηρότητες. Ε, το ανέλαβε το θέμα η FDD. Επίσης, κατάρτιση ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η προφορική ερώτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια του Ιανουαρίου του 2019. Επίσης, οργανώνουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Διεθνούς Οίκου των Γυναικών από τη Ρώμη. Σε ό,τι αφορά το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχετικό νομοθετικό πακέτο, με βάση το άρθρο 54, οι συντονιστέ αποφάσισαν να καταρτήσουν γνωμοδότηση για το πρόγραμμα ε, Δικαιώματα και Αξίες. Το αναθέσαμε στο ΕΛΚ. Επίσης, ε, πρόβλεψαν γνωμοδότηση για την κοινή γεωργική πολιτική που την ανέλαβε το ΕΛΚ. Επίσης, κατάρτιση γνωμοδότηση για το ενισχυμένο κοινωνικό ταμείο θα την ε, συντάξει το ΕΛΚ και έκθεση για το Μηχανισμό Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία. Ε, την ανέλαβε η ΓΚΟΕ. Επίση, ε, με τη μορφή τροπολογιών θα παρουσιάσουμε τη θέση μα στην έκθεση τη Επιτροπή Απασχόληση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Θα εκπονήσει το σχετικό σχέδιο η Πρόεδρος και επίσης γνωμοδότηση προς την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για την ε, θέσπιση του προγράμματος δικαιοσύνη κάτι που ανέλαβε ε, αρμόδιος από τους φιλελεύθερους. Περάμε στο σημείο 4, το πιο σημαντικό για σήμερα. Είναι η δημόσια ακρόαση για το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος. Στις 24 Ιανουαρίου του 2018, οι συντονιστές αποφάσισαν να διοργανώσουν δημόσια ακρόαση με θέμα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη διετία 2017-2019 με θέμα την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Ε, επίσης, ο ε, στόχος είναι η ανάλυση των προτάσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017-2019 και κυρίως η αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων, που είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη ζωή τους. Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλους τους οικονομικούς κλάδους, κερδίζουν κατά κανόνα 16% λιγότερο από ό,τι οι άντρες. Στην ακρόασή μας θα ακούσουμε τον Γενικό Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Προστασίας του Καταναλωτού, επίσης εκπροσώπους των εργοδοτών και εργοζομένων και εκπροσώπους ε, πανεπιστημίων. Το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο έχει την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων και την γεφύρωση αυτού του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Περνάμε τώρα στο πάνελ τη δημόσια ακρόαση. Θα ακούσουμε πρώτα τρεις καλεσμένους, καλεσμένες για την ακρίβεια, την Τίνα Άστολα, που είναι Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ε, για τη Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καλώς ήρθατε. Μετά τη Vivian Hunt, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της McKenzie Company, ε, Ηνωμένου Βασιλείου και και την Ingrid Moritz, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Γυναικών στο Αυστριακό Εργασιακό Επιμελητήριο. Αυτές θα είναι οι τρεις πρώτες καλεσμένες μας. Θα τις ακούσουμε για 10-15 λεπτά και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ με τις τρεις επόμενες εμπειρογνώμονες. Πρώτα λοιπόν θα ακούσουμε την κυρία Τίνα Αστόλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στη σημερινή ακρόαση να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Και για το σημερινό κοινό μας που βλέπω αποτελείται κυρίως από γυναίκες, ευτυχώς όχι όμως αποκλειστικά. Η μισθολογική ισότητα έχει θεσπιστεί ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και έκτοτε οι γυναίκες έχουν ε, εισέλθει μαζικά στην αγορά εργασίας, ωστόσο ε, βγάζουν ακόμα 60% λιγότερο κατά μέσο όρο από τους άντρες. 16%, 16% συγγνώμη. Και αυτό είναι ένδειξη της ανισότητας και αποτελεί και εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς. η προώθηση της ε, ίσης αμοιβή των γυναικών είναι κάτι από το οποίο μπορούν να κερδίσουν όλοι, είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη κοινωνία, είναι όμως και κίνητρο για οικονομική ανάπτυξη. Στις 20 Νοεμβρίου πέρσι, ο Επίτροπος υιοθέτησε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι αιτίες για το μισθολογικό χάσμα είναι πολυσχηδείς, προέρχονται από στερεότυπα, από ανεπαρκή επιβολή του νόμου και έλλειψη διαφάνειας. Υπάρχει λοιπόν ευρύ φάσμα αιτιών για το μισθολογικό χάσμα. Γι' αυτό χρειάζεται μείγμα πολιτικής και άλλων μέτρων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις. Απαιτείται προσήλωση αυτών που χαράσουν την πολιτική και σε, και σε ευρωπαϊκό και σε ε, εθνικό επίπεδο. Η αρχή της ίσης αμοιβή ε, θεσπίζεται στη συνθήκη και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί ε, κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ίση αμοιβή. Και επίσης ευαισθητοποιούμε διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες ε, σχετικά με την σωστή εφαρμογή των ισχυών των κανόνων. Υπάρχει ε, κάθετη αλλά και ε, οριζόντια απομόνωση σε κάποιους τομείς. Οι γυναίκες ε, ακόμη δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην ηγεσία, ενώ εισέρχονται με τις ίδιες προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας. Επίσης, συχνά διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους επειδή πρέπει να φροντίσουν κάποιο παιδί, για παράδειγμα. και ε, πληρώνουν ε, ένα δυσανάλογα υψηλό τίμημα γι' αυτό. Επίσης, οι συντάξει των γυναικών είναι 40% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών. Υπάρχει λοιπόν και η απειλή φτώχειας ε, στην τρίτη ηλικία για τις γυναίκες. Το σχέδιο δράσης εξετάζει διάφορους τρόπους καταπολέμησης των διαφορών αυτών θέλουμε να αμφισβητήσουμε τα στερεότυπα και καλούμε τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν, ε, για παράδειγμα, τις ε, ανεπαρκείς αμοιβέ στον ε, εκπαιδευτικό τομέα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε γυναίκες να εισέλθουν σε επαγγέλματα που συνήθως δεσπόζονται από τους άντρες, όπως είναι οι μεταφορές, ή αντιστρόφως τους άντρες σε γυναικεία επαγγέλματα. Άλλη δράση στόχο έχει να προωθήσει την ε, ισότητα στις αδειοδρομίες. Φέτος είχαμε πάνω από 100 αιτήσει ε, για βραβείο γυναικείας ε, καινοτομίας. 10 επιχειρήσεις μπήκαν στον τελικό, ενώ τρεις επιχειρηματίες από την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το διαδίκτυο των πραγμάτων και της κοινωνικής υπηρεσίας βραβεύτηκαν. Επίσης, όσον αφορά τον ε, κοινωνικό αποκλεισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη στην ε, ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και προωθεί σχετική πρόταση πριν τις επόμενες ευρωεκλογές. Επίσης, έχουμε μια πρόταση για την ε, εξισορρόπηση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, συμφωνήθηκε μια κοινή προσέγγιση και προσβλέπουμε στους τριμερείς διαλόγους για θέματα συνομοθεσίας και προσβλέπουμε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Η διαφάνεια στις αμοιβέ είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να ε, διαφωτιστούν οι ανισότητες εντός επιχειρήσεων. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση για την ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβή ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας. Η σύσταση αυτή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις για να εντοπίσουν ενδεχόμενα μισθολογικά χάσματα. Τα μέτρα αυτά λοιπόν επιτρέπουν σε άτομα να ζητήσουν πληροφορίες ε, σχετικά με το ύψος ε, αμοιβή ε, εργαζομένων και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποβάλουν εκθέσεις, να εφαρμόζουν λογιστικούς ελέγχους και άλλα μέτρα. Και μαζί με το σχέδιο δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης υιοθέτησε αξιολόγηση των στις 20 Νοεμβρίου σχετικά με την εφαρμογή αυτής της σύσταση. Τέσσερα χρόνια μετά από την υιοθέτηση της σύσταση αυτής, βλέπουμε ότι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μόλις το 1 τρίτο των κρατών μελών έχει υιοθετήσει νομοθετικά μέτρα για να αυξήσει την μισθολογική διαφάνεια. Η έλλειψη πρόοδου δείχνει την ανάγκη για πιο στοχευμένα μέτρα στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια. Αξιολογούμε λοιπόν τις διατάξεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στην οδηγία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Και αυτή είναι μία από τις δράσεις που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης. Το μισθολογικό χάσμα είναι και ένας από τους δείκτες που εμφανίζονται στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρακολούθηση του κοινωνικού πυλώνα και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως βλέπετε από τις ε, αναχώρα στάσεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Μάιο του 2018, το μισθολογικό χάσμα παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Το μεγάλο χάσμα συνεχίζει να είναι προβληματικό στην Αυστρία, την Εστονία, τη Γερμανία και το 2018 τέθηκε ως νέο θέμα ε, στην Τσεχία και την Σλοβακία. Είμαι Φιλανδή, δεν υπάρχει ε, σύσταση αναχώρα για τη Φιλανδία. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι συνεχίζει να είναι σημαντικό το μισθολογικό χάσμα, ενώ η Σουηδία είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς ως συνήθως. Η ισότητα των δύο φύλων είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή. Απομένουν πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γενική Διευθύντρια. Ευχαριστούμε και για τις προτάσεις και τις συστάσεις που μας κάνατε. ιδιαίτερα για τις προτάσεις περί διαφάνειας ε, των μισθών που ίσως είναι κάπως ε, επίμαχη, αμφιλεγόμενη λύση για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και φαντάζομαι αυτό θα προκύψει και από την παρέμβαση της επόμενης μας καλεσμένης, κυρίας Vivian Hunt. Παρακαλώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ τους βουλευτές, τη γραμματεία, την πρόεδρο, τους διερμηνείς και όλη την ομάδα για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα της στήριξης των δικαιωμάτων των γυναικών για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αλλά και το μισθολογικό χάσμα. Εδώ στην Ευρώπη ξεκίνησε η εταιρεία μας και στην Γαλλία πιο συγκεκριμένα ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την ισότητα των δύο φύλων και τώρα έχουμε πλέον α, επεκταθεί στην δύναμη της ισότητας, ένα θέμα που αφορά 192 χώρες και βέβαια στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις της α, ισότητας, της ίσης εκπροσώπησης των α, εργασιακό χώρο, της ίσης συμμετοχής αλλά και της εξάλληψη του μισθολογικού χάσματο. Ε, είναι τιμή μα λοιπόν που μιλάμε σήμερα εδώ και σα ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε ό,τι αφορά την αξία της ε, συμμετοχής των δύο φύλων είναι σημαντικό για την οικονομία και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ερευνητές μας βρίσκουν ότι αν καταφέρουμε να κλείσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα, αυτό θα μπορούσε να αποφέρει 22-3 εκατομμύρια στην οικονομία συνολικά απέναντι σε αυτήν την ε, πρόκληση οι διάφορες εταιρείε προσπαθούν να επιτύχουν το καλύτερο για την περιφερειά τους αλλά και για την ε, χώρα τους. Δοκιμάσαμε, κάναμε πειράματα στο Σαν Πάολο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και είδαμε ότι ακόμη και σε αυτά τα πρότυπα υπάρχουν τεράστιες, τεράστια κέρδη αν καταφέρουμε να κλείσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα της τάξης των 12-3 εκατομμυρίων. Ε, προτιμάμε έναν πιο ευέλικτο τρόπο εργασίας 20% των κερδών αυτών θα μπορούσε να επέλθει από γυναίκες που θα είναι σε καλύτερες θέσεις εργασίας και 20% από πιο ευέλικτα προγράμματα. Οι περισσότερε οικογένειε, τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν ανάγκη από μεγαλύτερο εισόδημα, έχουν ανάγκη από περισσότερη δουλειά. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα το πιθανό κέρδο θα μπορούσε να φτάσει τα 6,13 εκατομμύρια. Σε συγκεκριμένε περιφέρειες θα μπορούσε να φτάσει το 2, τα 2,13 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτό το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος και στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Κατά τη γνώμη μας, η απάντηση περιλαμβάνει δύο στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει με τους τομείς που είναι η πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην οικονομία, η πιο παραγωγική. Ο τομέα τη ενέργεια, των μετακινήσεων, ο χρηματοοικονομικό τομέα, ο τομέα τη υγεία. Όλα αυτά είναι παραδείγματα τομέων που είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί. Άλλοι τομεί είναι η γεωργία κτλ. που μπορεί να έχουν χαμηλότερη παραγωγικότητα. Καταλαβαίνοντα όμω πού βρίσκονται οι γυναίκε, πού εργάζονται και σε ένα ιδανικό σενάριο να, τους έχουμε, να, να τις έχουμε να δουλεύουν σε πιο παραγωγικούς τομείς θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο δεύτερος παράγων που θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση του μισθολογικού χάσματος είναι αυτή η ιδέα της προαγωγής στον ε, ιδιωτικό τομέα, ε, το να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους το να έχουμε γυναίκες σε υψηλότερες θέσεις εργασίας, είτε ως ε, διευθύντριες, είτε σε ηγετικέ θέσεις, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ισότητα, αλλά και στο κλείσιμο του μεσολογικού χάσματος. Εδώ στο παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο που βλέπετε, αυτό που κοιτάμε είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι γυναίκες συνήθως βρίσκονται σε χαμηλότερα παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και σε λιγότερο ηγετικέ θέσεις. Και ο συνδυασμός των δύο αυτών ε, παραγόντων οδηγεί και στο μισθολογικό χάσμα. Οι άντρε αντιθέτως βρίσκονται σε ε, υψηλότερους ε, παραγωγικά τομείς και σε υψηλότερες θέσεις. Η διαφάνεια λοιπόν σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ, σύμφωνα με τον νόμο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νόμος που ξεκίνησε από την άνοιξη αυτού του, του χρόνου και ζητήσαμε από πάρα πολλές εταιρείες να μας αποκαλύψουν τις αμοιβέ των υπαλλήλων. Αν δούμε τα νούμερα, αυτό που είναι ανάγκη να κάνουμε είναι το εξής. Να βάλουμε γυναίκες σε, πιο, σε παραγωγικά αυξημένους τομείς, αλλά και σε πιο ηγετικές θέσεις. Εξετάζοντας λοιπόν και εισάγοντα του δύο αυτούς τομεί στο σχέδιο δράσης, θα μπορούσαμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο ιδιωτικό όσο και ο δημόσιο τομέα μπορούν να κάνουν πολλά για να κλείσουν το μισθολογικό χάσμα. Η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνηση. Στη συνέχεια όμω αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε στοχευμένε, ολοκληρωμένε παρεμβάσει σε βάθο χρόνου. Ιδίω καθώ έχουμε εκλογέ, όπω ξέρει η Κομισιόν, και θα πρέπει η νέα επιτροπή να δεσμευτεί διότι τα οικονομικά ωφέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά για τι γυναίκες αλλά και για την οικονομία συνολικά. Είναι ανάγκη όμως να έχουμε συντονισμένες προσπάθειες σε βάθος χρόνου. Κίνητρα, αλλά και ενθάρρυνση, καλύτερη τεχνολογία για την ε, διαφάνεια, συγκεκριμένες οικονομικές προοπτικές για, να, για ανάπτυξη, βοήθεια, συστηματική παρακολούθηση να βλέπουμε κατά πόσο σημειώνεται πρόεδρος και βεβαίως κανόνες και κανονισμούς που μπορούν να στηρίξουν α, αυτού του τύπου την πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της, του μισθολογικού χάσματος και της ισότητας, είναι μια συζήτηση που βρίσκεται στην επικαιρότητα και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποβάλουμε ολοκληρωτικά τα διάφορα στερεότυπα γνωρίζουμε ότι 75% των γυναικών που είτε εργάζονται τώρα είτε θα ήθελαν να εργαστούν θα έχουν θετικές επιπτώσεις από αυτού του τύπου τις πολιτικές. Και πάλι όμως έχουμε ανάγκη από συστηματικές παρεμβάσεις. Ξέρουμε ότι το τίμημα αξίζει. οι εταιρείε που έχουν μεγαλύτερη ποικιλία, μεγαλύτερη ε, στα, στα, σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους τους, έχουν καλύτερες επιδόσεις, η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη φτάνει το 21% και σε ό,τι αφορά την δημιουργία προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 27% μεταξύ των εταιριών που έχουν μεγαλύτερη ποικιλία σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλου τους. Τρία θέματα θέλουμε να σας δώσουμε. Είναι δυνατή η πρόοδος. Μπορούμε να προοδεύσουμε σε ό,τι αφορά το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος με το να βάζουμε γυναίκες σε παραγωγικά δυνατούς τομείς, αλλά και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ε, υψηλές, όπου συμβάλλουν στην ε, διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Δευτερευόντως, πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο για να ενδυναμώσουμε την νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορούν την διαφάνεια όταν οι επενδυτές αλλά και οι κοινωνίες οι ίδιες δουν ποια είναι η αξία, τότε θα είναι οι ίδιοι διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε πάνω στην ιδέα της αλλαγής του εργασιακού περιβάλλοντος. Η τεχνολογία και πολλοί άλλοι παράγοντες αλλάζουν ολοσχερό στο περιβάλλον της εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια φρέσκια αρχή, να μην επαναλάβουμε αυτά τα ίδια στερεότυπα που αφορούν τις γυναίκες. Είναι ανάγκη να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην υψηλή τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς. και κυρίως το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες σε αυτόν τον χώρο της τεχνολογίας. Διατρέχουμε τον κίνδυνο και σε αυτή τη νέα οικονομία να επαναλάβουμε και πάλι τα στερεότυπα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Είναι λοιπόν ανάγκη να σκεφτούμε εκ των προτέρων και στο χτίσιμο αυτής της νέας οικονομίας να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τη νέα θέση της γυναίκας ούτως ώστε να επιτύχουμε και την ταχύτερη ανάπτυξη από κοινού μαζί με, τη, με το σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. And, uh, Και περνάμε τώρα στην τρίτη μας καλεσμένη, την Ingrid Moritz, επικεφαλής του Τμήματος Γυναικών του Αυστριακού Εργατικού ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω την παρουσίασή μου στα γερμανικά γιατί είναι πιο εύκολο για μένα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάχω στη σημερινή ακρόαση. Ε, το Αυστριακό επιμελητήριο Εργασίας ε, είναι μια ένωση για όλους τους επιχειρηματίες ε, της Αυστρίας. 3,7 εκατομμύρια μέλη έχουμε και μας ενδιαφέρει η πολιτική για τους εργαζομένους, οι βάσεις για την εργασία, παρέχουμε σύμβουλες και ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρει είναι η μισθολογική δικαιοσύνη. Θέλουμε να κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα και ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων. Εδώ και πολλά χρόνια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται στατιστικές ε, για να φανεί πόσο μεγάλο είναι το μισθολογικό χάσμα και για να δοθούν κίνητρα για περισσότερη μισθολογική δικαιοσύνη. Η ιεράρχηση δείχνει ότι η Αυστρία ήταν εδώ και πολλά χρόνια στην πρώτη-τελευταία θέση. Πολύ σημαντικό επίσης ήταν ο στόχος της Βαρκελόνης όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών. Με αυτό καταφέραμε στην Αυστρία να δώσουμε κίνητρα για καλύτερη φροντίδα των παιδιών για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. αναφέρονται οι στόχοι που θέλει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό όμως είναι και η υποβολή εκθέσεων και η καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού. Το μισθολογικό χάσμα στην Αυστρία αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 21,7%, μεγαλύτερο δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν ο τελευταίος τροχός της ε, αμάξης και το 2011 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις

που καλύπτονται από τις ε, συλλογικές ε, συμβάσεις, ε, καθώς και η αμοιβή τους. Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται με ανωνυμοποιημένη μορφή. Δεν υπάρχει κύρωση σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η έκθεση αυτή. Το Συμβούλιο εργασία όμως μπορεί να ζητήσει μέσω δικαστηρίου την εκπόνηση της έκθεση. οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν συμβουλές από ε, τις οργανώσεις στις οποίες ανήκουν, για παράδειγμα και ε, από το Αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας. Συμπεράσματα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εκπονούν την έκθεση αυτή, μόλις όμως το 26% των εργαζομένων γνωρίζουν την ύπαρξη της έκθεσης αυτής. Σε πολλές επιχειρήσεις με τις μισθολογικές αυτές εκθέσεις. Ε, υπάρχει συστηματική επισκόπηση των ε, μισθών, κάτι που δεν ίσχυε πριν ε, και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο επαγγελματισμό όσον αφορά την πολιτική αμοιβών. Αναθέσαμε την εκπόνηση γνωμοδότησης και τα συμπεράσματα. δείχνουν ότι όταν υπάρχει υποψία μισθολογικής διάκρισης, αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί με τη δικαιολογία των ε, ε, επαγγελματικών εμπιστευτικών πληροφοριών. Πολύ Επίσης, οι ρήτρε ε, που λένε ότι δεν επιτρέπεται να ε, αναφέρει κανείς ε, ποια είναι η αμοιβή του, απαγορεύονται πια. Επίσης, όσον αφορά δημόσιες συμβάσεις καθώς και εσωτερικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών, έχουν αλλάξει οι κανόνες. Και Τα συμπεράσματα από τους ε, νέους κανόνες ε, είναι ότι επειδή δεν υπήρξε κύρωση, δεν εφαρμόστηκαν οι νέοι κανόνες, ε, μόνο μετά την επιβολή κύρωσης τηρήθηκαν οι κανόνες. Συχνά όμως αναφέρεται μόνο η ελάχιστη αμοιβή σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις. το 44% των εργαζομένων πιστεύουν ε, ότι οι άντρες ε, αναφέρουν ότι λαμβάνουν μεγαλύτερο μισθό όταν ε, δεν είναι απαραίτητο να υποβάλει κανείς το ελάχιστο. Είναι σημαντικό εργαλείο αυτό για την αυτοαξιολόγηση των γυναικών απομένουν πολλά να γίνουν, διότι ακόμη βλέπουμε ότι ελάχιστες υποθέσεις ε, για μισθολογική διάκριση καταλήγουν στο δικαστήριο, ενώ η ψαλίδα ε, είναι πολύ μεγάλη. Ζητάμε λοιπόν απόλυτη μισθολογική διαφάνεια, ώστε να μπορεί κανείς ε, πραγματικά να συγκρίνει την αμοιβή του με αυτήν των συναδέρφων. Η εκθέσεις, οι μισθολογικές δεν θα πρέπει απλά να υποβάλλονται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και ως βάση για μείωση της μισθολογικής ψαλίδας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον συνδυασμό ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, που είναι πολύ σημαντικό παράγοντα για το μισθολογικό χάσμα. Βλέπουμε ότι οι ώρες εργασίας, για παράδειγμα, δυσκολεύουν ε, την κατάσταση για πολλές γυναίκες. Επίσης, κάθε... με κάθε ε, ώρα εργασίας του άντρα πέρα από την κανονική ώρα εργασίας ε, αυξάνεται το μισθολογικό χάσμα. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος να γίνει πιο δύσκολο ο συνδυασμό επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, κάτι που θα δυσκολέψει τα πράγματα ακόμα περισσότερο για πολλές γυναίκες και έτσι θα αυξηθεί το μισθολογικό χάσμα. Θα είναι σημαντικό να συζητηθεί αυτό το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία παρατήρηση. όσον αφορά τις ε, ρήτρες σε μία αναστρεψιμότητας στις οδηγίες που υπάρχει στην ε, οδηγία για τον ε, συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου και σημαντικό είναι να μην υπάρχει αναστρεψιμότητα. Στην Αυστρία γίνεται αυτή τη στιγμή ε, το θέμα του gold plating, του να είναι πιο αυστηροί οι εθνικοί κανόνες ε, από τους ευρωπαϊκούς. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σωστές διατάξεις στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Thank all... Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις τρεις καλεσμένες μας, την, την Άστολα, την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Vivian Hunt από τη McKenzie Company, από τη του Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδία και την κυρία Μόριτσα, ε, Διευθύντρια του Τμήματο Γυναικών του Αυστριακού Εργατικού Επιμελητηρίου. Περνάμε τώρα στι τρεις επόμενες καλεσμένε. Ε, στην κυρία από την Deloitte, Τμήμα Αναζήτηση Ταμείων, ε, τη Γενική Διευθύντρια Καθρίνα, Καθρίνα Μίλλερ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών Δικηγόρων. Θα ήθελα να καλέσω τις τρεις επόμενες εμπειρογνώμονες να λάβουν το λόγο να καθίσουν στο πάνελ. Okay, so the... Μάλιστα. Το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης ήταν πολύ ενδιαφέρον και προκάλεσε πολλές ερωτήσεις, αλλά πρώτα θα ακούσουμε τις άλλες τρεις καλεσμένες, ώστε να ολοκληρώσουμε τις παρουσιάσεις από τους εμπειρογνώμονες και θα περάσουμε στην κυρία Έμα Κότ, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος ε, στο Τμήμα Ταλέντων τη Deloitte του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε καταρχήν. Θα σας μιλήσω καταρχήν για το ταξίδι που κάναμε εμείς στην Deloitte του Ηνωμένου Βασιλείου την τελευταία τετραετία. Στην πορεία μας αυτή την τελευταία τετραετία. Μου ζήτησαν να σας παρουσιάσω πώς εμείς ως οργάνωση καταφέραμε κάποιες ουσιώδεις αλλαγές, ποιο ήταν το ταξίδι που κάναμε, ποια η πορεία μας, ε, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα αποτελέσματα. Εγώ, ε, ω διευθύνων σύμβολο για τα ταλέντα, μου δίνει την ευθύνη για ό,τι κάνουμε για του 16.000 ε, μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίση ε, έχουμε 34.000 συνολικά από την βόρειο-δυτική Ευρώπη, αλλά σήμερα θα επικεντρωθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας ε, επαναφέρω στο 2012 και ο λόγος που το κάνω είναι ότι τότε, το 2012, κάναμε μια πολύ γενναία, θαραλέα τότε κίνηση και θέσαμε κάποιους στόχους για την εκπροσώπηση των φύλων στα πιο υψηλό βαθματιμάτα της ε, οργάνωσής μας, σε επίπεδο των συμβούλων δηλαδή. Ε, τότε είχαμε μόνο 12% των εταίρων μας σε διοικητικέ, υψηλές διοικητικές θέσεις που ήταν γυναίκες και αποφασίσαμε αν κάτι ήταν σημαντικό για μα. θα έπρεπε όχι μόνο να θέσουμε στόχους, ε, να συντάξουμε ένα δημοσιονομικό ε, σχέδιο και άλλα ε, οικονομικά ζητήματα που ήταν σημαντικά, αλλά να καταμετρήσουμε και τη μέθοδο και την πρόοδο υλοποίηση των στόχων. Το 2013 διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ακόμη πρόοδος. Μόνο 12% των εταίρων μας, ε, των διευθυντικών μας ε, μελών ήταν γυναίκες. Οπότε ε, καθίσαμε μαζί με τα άλλα στελέχη και αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση για να επιφέρουμε πραγματικά ουσιώδεις αλλαγές. Τελικά κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι οργανώσεις. Εξετάσαμε πρώτα τα δεδομένα μας και τα δεδομένα μας μας έδειξαν πολύ στερεότυπα στοιχεία. Για παράδειγμα, όλες οι οργανώσεις θέλουν να λένε ότι έχουν 5% εκπροσώπηση των φύλων στο σημείο εισόδου. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Μέσα σε μία δεκαετία είχαμε από 50% στο 36% μείωση. Άρα ξεκινήσαμε από πολύ κακή αφετηρία. Και αν δει κανείς ολόκληρη τη σταδιοδρομία των μελών, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες που ήταν επιτυχημένε κατά τη στιγμή της πρόσληψης, παρέμεναν στην εταιρεία 6 με 8 χρόνια. Και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα είχαν μία ε, απομάκρυση από τις ε, ε, ηγετικές θέσεις. Και ποιος ήταν ο λόγος. Καταρχήν είδα, οι γυναίκες έβλεπαν ότι οι συνάδελφοι τους άνδρες προαγόνται με ταχύτερους ρυθμούς ή άλλες γυναίκες ασχολήθηκαν με την οικογένειά τους ή άλλα μέλη της οικογένειας που έπρεπε να φροντίσουν ήταν να μεγαλώσουν παιδιά. Και μάλιστα όταν επέστρεφαν στην αγορά εργασία, ε, διαπίστωναν ότι δεν μπορούν να συνδυάσουν τον προσωπικό με τον επαγγελματικό βήλο. Επίση, είδαμε ότι η θωρά των γυναικών ε, ήταν πολύ πιο μεγάλη από των ανδρών. Επίση, είδαμε ότι δεν ήταν τόσο ενθουσιώδει οι γυναίκε, οι προσιλωμένε στη δουλειά όπω οι άντρε. Και ε, διαπιστώσαμε με του εταίρου ότι δεν ήταν μόνο στην εταιρεία μα αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε πολλέ υπηρεσίε υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Οπότε έπρεπε να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα. Συναντηθήκαμε με τις ε, γυναίκες της εταιρεία και τις ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουμε για να παραμείνετε στην εταιρεία, για να μας επιλέξετε, για να συνεχίσετε τη σταδιοδρομία σας. Και μας είπαν ξεκάθαρα τι ήθελαν. Ε, ήθελαν να νιώθουν ότι προόδευαν, ε, πρόκοβαν στη σταδιοδρομία τους, αντίστοιχα με τους άνδρες. Και κυρίως μας είπαν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην κουλτούρα της εταιρεία. Και όταν μιλήσαμε για την κουλτούρα της εταιρεία, σταθήκαμε σε δύο κυρίως σημεία. Ε, συμφιλίωση του προσωπικού με τον επαγγελματικό βίο. Είχαμε ε, ευέλικτες μορφές εργασίας, αλλά όχι αρκετά προσιτές. Επίσης, αυτό που στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάποια σχόλια που γίνονται ε, εν είδη αστείο συναδέλφους, που δεν είναι καθόλου όμως ε, αστείες και σταδιακά επηρεάζουν τη σταδιοδρομία των γυναικών και υπονομεύουν την ε, αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη των γυναικών και την πίστη τους προς τον οργοδότη τους. Οπότε σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο δράση και μάλιστα ήμασταν ξεκάθαροι γι' αυτό μαζί με τους διευθύνοντες, συμβουλίους, ε, διευθύνοντες συμβούλους. Ε, και μάλιστα σκεφτήκαμε ότι το θέμα δεν θα έπρεπε να το αναλάβει το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, αλλά η διεύθυνση. Και δημοσιεύσαμε το σχέδιο το σχέδιο δράσης ε, χωρίς ντροπή γιατί θέλαμε όλοι να αντιληφθούν ότι είχαμε επιθυμία και σκοπό να κάνουμε ουσιαστικές και ρεξικέλευτες αλλαγές. Έπρεπε πρώτα να, ξεκινά, να τροποποιήσουμε την κουλτούρα της εταιρεία. Καταρχήν, ε, όταν ρώτησα την ομάδα μου γιατί έχει μειωθεί στο 36% η, προσλήψη, η προσλήψη των γυναικών μου, ε, είπαν οι διευθύνοντες ότι περισσότερο ζητούσαμε δεξιότητες σε θετικές επιστήμες. και οι γυναίκες δεν προτιμούν τόσο τις θετικές επιστήμες. Επίσης, ε, είδαμε τη διατύπωση που χρησιμοποιούσαμε. Χρησιμοποιούσαμε ούτως ή άλλως ένα λεξιλόγιο που απηχούσε περισσότερο σε άνδρες. Δεν ήταν τόσο ελκυστικό για τις γυναίκες που θέλαμε να προσελκύσουμε στην οργάνωσή μας. Επίσης, υπήρχαν και άλλα, άλλα στοιχεία. Όταν κοιτάζουμε το σύστημά μας, όταν βλέπουμε το πώς προσπαθούσαμε να συνεργαστούμε με τις γυναίκες για να τις προσελκύσουμε στην οργάνωση, διαπιστώσαμε ότι η ίδια μας η διαδικασία ήταν το πρόβλημα. Γιατί ε, εφαρμόζαμε τη σειρά προτεραιότητες. Οι γυναίκες ναι μεν εξέφραζαν ενδιαφέρον, αλλά μετά άρχισαν να το σκέφτονται. Ε, για το αν στεριζόμαστε τις ίδιες αξίες ε, και στο μεταξύ όταν λάβανα την απόφαση και, εμείς, και επέστρεφαν εμείς είχαμε ήδη κάνει τις προσλήψεις. Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη χαμηλή πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις, είχαμε κάποιες παρεμβάσεις, ε, κάποια προγράμματα προ, κατά κάποιο τρόπο mentoring για τις γυναίκες. Επίσης, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουν οι γυναίκες να συνεργαστούμε μαζί τους, να έχουν τους κατάλληλους χορηγούς για να μπορέσουν να αναδείξουν το δυναμικό τους. Επίσης, έχουμε μια πολύ σαφή ε, ιδέα τώρα τα τελευταία έξι χρόνια και τις προωθούμε σε πιο ηγετικές θέσεις. Επίσης, το θέμα το μισθολογικό. Θα έρθω σε αυτό αργότερα. Πάντως, τίποτα από αυτά που κάναμε δεν ήταν ε, μια προσπάθεια να διορθώσουμε τις γυναίκες. Αυτό που έπρεπε να διορθώσουμε ήταν ο χώρος εργασίας. Ε, χρειαζόμαστε ένα εξυγχρονισμό, μια κατάρριψη των ε, φραγμών και των εμποδίων που είχαμε συγκεντρώσει κατά την μακροχρόνια πορεία μας, των 150 χρόνια. Επίσης έπρεπε να καταμετρήσουμε την πρόοδο και να δούμε ότι όντως υπήρξε διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Καταρχήν ως προς την ευέλικτη εργασία. Το όρο ευέλικτος βέβαια το καταργήσαμε, το αντικαταστήσαμε το σβέλτος. Σβέλτος που είναι κάτι θετικό, κάτι ε, καλό και δίνει την ευκαιρία σε όλους και άνδρες και γυναίκες να εξασφαλίσουν αυτή την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μέσω διαρθρωμένων προγραμμάτων. Και το μυστικό της επιτυχίας μας ήταν η αλλαγή της κουλτούρας της οργάνωσης. Και δεν θα ήθελα να να υποτιμήσουμε τη σημασία που έχει αυτή η αλλαγή της κουλτούρας. Γιατί πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνονται την ευελιξία, αλλά δεν τη διαλέγουν μερικές φορές για να μην κατακριθούν από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Εμείς πραγματικά επικεντρώσαμε σε αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας της κουλτούρας. ό,τι αφορά την συμπερίληψη, ε, σκεφτήκαμε ότι χωρίς συμπερίληψη, χωρίς σεβασμό δεν θα έχουμε και πολυμορφία στην εκπροσώπηση. Και φυσικά για όλα αυτά χρειαζόταν και αλλαγή της νοοτροπίας. Και 6.000 από, τους, ε, από τα μέλη μας τα συμπεριλάβαμε σε προγράμματα κατάρτισης και είπαμε στον κόσμο πόσα προσόντα έχει. Προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε, να τους εψυχώσουμε και να τα προωθήσουμε καλύτερα. Επίσης είχαμε συμβούλους για την συμπερίληψη με κατάλληλους τρόπους ε, για ευαισθητοποίηση γιατί όταν ρωτήσαμε ε, τα μέλη αν έχετε προβλήματα, γιατί δεν αποτείνεστε στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων. Και όλοι μας είπαν, μα γιατί δεν τα παίρνουν αρκετά στα σοβαρά ή δεν θέλω στον προϊστάμενό μου να κάνω ένα επίσημο παράπονο. Οπότε εμεί δημιουργήσαμε διάβλους για την υποβολή τέτοιων παραπώνων και αλλάξαμε την οτροπία ολόκληρη. Οπότε τρία χρόνια μετά τι γίνεται. 50% αύξηση των ε, ε, εταίρων. Ε, των διεθνών των εταίρων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο στόχο, αλλά υπάρχει μια σημαντική πρόοδος. Επίσης, πρόσληψη φοιτητών είναι 45%. Ε, Δεν έχουμε φτάσει ακόμη το 50%, αλλά έχουμε βελτιώσει την τελευταία διετία κατά πολύ το ποσοστό. Επίσης, για τα ηγετικά στελέχη, έχουμε ε, αρκετές γυναίκες πια σε ηγετικές θέσεις. Δεν έχουμε τόση φθορά όσο στο παρελθόν και έχουμε πολλές γυναίκες που εργάζονται με τέτοιο ελαστικό τρόπο. Επίσης, έχουμε ένα καταπληκτικό σχέδιο εφαρμογής και γιατί κερδίσαμε. Κερδίσαμε αργά αλλά σταθερά. Γιατί είχαμε στόχους, είχαμε τρόπο καταμέτρησης των στόχων και της πρόοδου. Γιατί το θέμα δεν είναι έχουμε μόνο στόχους, αλλά και να μπορούμε να τους αξιολογούμε. Επίσης, λογοδοσία των ηγετικών στελεχών άνοιγμα και διαφάνεια. Έχουμε πολλή εκθέσεων για, το, για τις μισθολογικές ε, διακρίσεις. Από το 2015 εμείς οικειοθελώς συμμετέχουμε σε αυτή την απογραφή, ε, την καταγραφή μάλλον των μισθολογικών διακρίσεων για να φαίνονται τα αποτελέσματα. Πρόοδος στην οτροπία, στην κουλτούρα. Τα προγράμματα είναι καλά, αλλά δεν θα έχουν ουσιώδη ε, επίδραση αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, αν δεν εξυγχρονιστεί η νοοτροπία. Επίσης, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ηγετικά στελέχη θα πρέπει να φουγκραστούν τις γυναίκες. Αυτό κάναμε, ακούσαμε τις γυναίκες, αναλάβαμε δράση, εντοπίσαμε τα προβλήματα στον τρόπο εργασίας, στις συμπεριφορές, στην αντίληψη. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ε, οι γυναίκες, δεν έπρεπε τις γυναίκες να διορθωθούν, αλλά η κατάσταση να διορθωθούν. Και είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που επιτελέσαμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η προοπτική που μας παρουσιάσατε. Και συγχαρητήρια. Μπράβο σας για την επιτυχία σας. Και τώρα το λόγο η κυρία Κλώη Σαμπρό, που είναι διευθυντρία της εκστρατείας για την ισότητα των φύλων στην ε, οργάνωση Business in the Community. Χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ να σας παρουσιάσω τη δουλειά που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και να σας εξηγήσω και τι έχουμε κάνει εμείς στην εταιρεία επιχείρηση για την κοινότητα. Να σας πω λίγο δύο λόγια για το ποιοι είμαστε. Είμαστε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι εδώ που βρίσκονται και εργάζονται για την ισότητα των γυναικών Είμαστε μια πολύ ιδιαίτερη εταιρεία. Προσπαθούμε να προωθήσουμε το μοντέλο των υπεύθυνων επιχειρήσεων όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνων και αυτό είναι ένα ευρύτατο θέμα όπως καταλαβαίνετε. Θα σας δείξω με λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε από κοινού με αυτούς που χαράζουν τις πολιτικές, προσπαθούμε να τους επηρεάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Έχουμε πολλές έρευνες και πολλές καμπάνιες ούτως ώστε να τους ενημερώνουμε. Συλλέγουμε λοιπόν δεδομένα ούτως ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα, μεταξύ άλλων. Γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε συστάσεις. Δημοσιεύουμε τις έρευνές μας επίσης, ούτως ώστε να είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, είμαστε κατά κάποιο τρόπο μια συμβουλευτική εταιρεία, και δεν θα έλεγα ότι είμαστε αποκλειστικά αυτό, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όμως επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, αναφορές που πρέπει να κάνουν για α, τις αμοιβέ των υπαλλήλων και τα λοιπά. Ιδού λοιπόν ο χάρτης της εταιρεία μας τον βλέπετε στην οθόνη. Η ευθύνη των εταιριών δεν περιορίζεται μόνο στο περιβάλλον και από εκεί που έρχομαι εγώ τουλάχιστον έχει να κάνει και με την διαφορετικότητα και τον μη αποκλεισμό. Ε, α, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ισότητα μεταξύ των φύλων, η φιλετική ισότητα αλλά και η ισότητα στις διάφορες ηλικίε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο με το μισθολογικό χάσμα. Ο τρόπος που υπολογίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαφορετικός από τα νούμερα που μπορεί να έχετε δει σε διάφορους ε, διαδικτυακούς τόπους. Βασικά, όταν μιλάμε για αναφορές του μισθολογικού χάσματος, μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό από τις ίσες αμοιβέ. Θα σας πω δύο λόγια γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ των ίσων αμοιβών και του μισθολογικού χάσματο. Οι ίσε αμοιβέ έχουν να κάνουν μεταξύ δύο ατόμων ή δύο ομάδε ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά φύλλα, βρίσκονται στην ίδια επαγγελματική θέση και δεν κερδίζουν τα ίδια χρήματα. Όταν ο ένα είναι γυναίκα και ο άλλο είναι άντρα, η γυναίκα παίρνει λιγότερα χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι η αμοιβή είναι άνηση. Είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ένας από τους παράγοντες του μισθολογικού χάσματος, αλλά όχι ο μοναδικός. Σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα τώρα, έχουμε να κάνουμε μεταξύ μια, μιας ομάδας γυναικών και μιας ομάδας ανδρών σε μια οργάνωση, σε μια χώρα και υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στο μισθολογικό χάσμα. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι οι άνισες αμοιβέ, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός. Δεν θα αναφερθώ στο επιχειρησιακό, στην υπόθεση των επιχειρήσεων, γιατί η Vivian το έκανε πριν από μένα. Ξεκινήσαμε με εθελοντικέ αναφορές, όπως σας ανέφερε και η ΕΕΜΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο πέντε επιχειρήσεις κάνουν τέτοιες αναφορές μετά από πέντε χρόνια. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι αυτή η εθελοντική αναφορά δεν αρκεί. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή μία νομοθεσία στην οποία έχουμε συμβάλει τα μάλα, ε, συμβουλεύουμε την κυβέρνηση, έχουμε αναλάβει ένα γενικό συμβουλευτικό ρόλο και είμαστε της άποψης ότι δεν θα πρέπει απλώς να δημοσιεύεται το μισθολογικό χάσμα, αλλά να βλέπουμε και τις διαφορές στα μπόνους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και να καταγράφουμε βεβαίως και την πρόοδο στον χώρο της εργασίας. Πρέπει να κρατάμε κατά νου ότι όταν μιλάμε για το μισθολογικό χάσμα δεν αρκεί για να περιγράψουμε την καθημερινή πραγματικότητα της ζωής όλων των γυναικών. Αυτό που συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει να κάνει αφορά 250 επιχειρήσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά τα, τα, χάσματα στις αμοιβέ και στα μπόνους, αυτό που είδαμε είναι ότι οι γυναίκες, καθώς αυξάνουν οι μισθοί, οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άνδρες. Αυτές οι αναφορές πρέπει να δημοσιεύονται κάθε χρόνο. Θα πρέπει να μπορεί κανείς να βρει τα στοιχεία αυτά, γιατί είδαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείε τα κρύβουν αυτά τα στοιχεία με έγγραφα PDF κτλ. Θα πρέπει να είναι εύκολο να αναζητήσει κανείς τα έγγραφα αυτά και να τα βρίσκει στα website των διαφόρων εταιριών. Πώς εξηγούμε το, το χάσμα, το σχέδιο δράσης αυτό είναι επιλογής, δεν είναι υποχρεωτικό. Πολλά όμως από τα μέλη επιχειρήσεις το έκανα. Να σας δώσω μια εικόνα, ρίξτε μια ματιά εδώ στην οθόνη. Πηγαίνει στην σελίδα της εταιρεία, πηγαίνει μάλλον στην ανάλογη ιστοσελίδα, πληκτρολογείς το όνομα της εταιρεία και κάθε εταιρεία ε, θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία για όλες τις νομικές οντότητες. Σε πολλές περιπτώσεις ε, διαθέτουν παραπάνω από μία νομική οντότητα οι εταιρείε μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορα φίλτρα και να ε, έχεις ένα αποτέλεσμα πιο συγκεκριμένο. Έβαλα ένα ερωτηματικό. Είναι επιτυχέ. Εγώ προσωπικά πιστεύω γιατί, ότι είναι επιτυχέ, γιατί 10.000 εργοδότες έκαναν αυτή την αναφορά. 99,9% ο βαθμός συμμόρφωσης. Γνωρίζουμε ότι επισκέπτονται τη σελίδα 9.000 φορές την ημέρα και όταν πρώτο ξεκίνησε υπήρξαν ε, πάρα μα πάρα πολλά hits, οι γυναίκες το χρησιμοποιούν. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά λάθη ε, στις αναφορές, για παράδειγμα κάποιες εταιρείες ε, σημειώνουν 0% μισολογικό χάσμα, το οποίο είναι αδύνατον. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζει αυτούς τους εργοδότες. Αυτό όμως το οποίο γίνεται και συζητάμε με τους εργοδότες που είναι μέλη της κοινότητάς μας, συζητάμε με εταιρείες που δεν είχαν επίγνωση του προβλήματος αυτός και τους εξηγούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι ανάγκη να δώσουμε έμφαση στο πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο να το εξηγήσουμε, αλλά να κάνουμε και κάτι. Έχουμε αρκετούς λοιπόν εταίρους ε, της ε, δικής μας οργάνωσης που μας ρωτάνε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να καταπολεμήσουν το πρόβλημα αυτό. Τι κάνουμε εμείς ως ε, επιχειρήσεις για τις κοινότητες. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τις γυναίκες είναι το να κάνουν παιδιά. Και αυτό που είδαμε με χαρά μου ήταν ότι υπάρχει ένα, μια κύρωση, η οποία δεν ονομάζεται κύρωση για τις μητέρες, αλλά για αυτούς, για τα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά. Care penalty και όχι mother penalty αν ε, ρίξετε μια ματιά στα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά, ανέρχονται σε 42%. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, μάλλον, θα έλεγα. Και θα έλεγα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά στα άτομα που δουλεύουν full time, δουλεύουν πολύ περισσότερο και οι γυναίκες δουλεύουν part time πολύ περισσότερο από σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό γιατί η φροντίδα των παιδιών είναι τόσο ακριβή, όπου οι γυναίκες αναγκάζονται να δίνουν μεγάλο μέρος του μισθού τους για την φροντίδα των παιδιών. Και είμαστε στη διαδικασία σύνταξης μιας αναφοράς, μιας έκθεσης, την οποία κάναμε από κοινού με μια εταιρεία ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί και με την αίμα που είναι εδώ σήμερα. Ζητήσαμε από 10.000 άντρε, τι πρέπει να γίνει διαφορετικά. Αν δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο του άντρε και στο σπίτι, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία και στις γυναίκε να βρίσκονται στο χώρο εργασία, Γιατί θα πρέπει να είναι πάντοτε οι γυναίκε που πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά, γιατί θα πρέπει οι γυναίκε να δουλεύουν αποκλειστικά part-time. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ε, δουλειά την καθημερινή, αλλά και σε ό,τι αφορά την, ε, συντάξει του. Um, Κάναμε λοιπόν μια πολύ εκτεταμένη έρευνα με διάφορους ακαδημαϊκούς ανεξάρτητους. Υπάρχει ένα βίντεο, αν έχουμε χρόνο να το δούμε. Ε, για καλό και για κακό θέλω να κλείσω τη συζήτηση αυτή. Η διαφάνεια, όπως είπε και η άμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Όταν οι ίδιες οι εταιρείες αρχίσουν να μετράνε, θα δουν ότι δεν μπορούν να, να κρυφτούν και μπορούν, θα πρέπει να λάβουν μέτρα δεν αρχεί να λέμε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να διαπραγματεύονται περισσότερο, το να διορθώνουμε τις γυναίκες. Αυτή είναι η λάθος ε, προσέγγιση. Έχουμε συνειδητοποιήσει μέσω πολλών ερευνών εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες. Δεν είναι πρόβλημα έλλειψη αυτοπεποίθησης ή, ή έλλειψης φιλοδοξίας. Είναι πρόβλημα του εργασιακού χώρου, είναι πρόβλημα διακρίσεων σε πολλές περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε αυτά τα προγράμματα, τα πιο, τα πιο ευέλικτα, τα πιο προσαρμόσιμα και βεβαίως να αποθαρρύνουμε τα πιο μη ευέλικτα συστήματα που δεν είναι καλά και για την παραγωγικότητα ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε να μοιράζεται η φροντίδα των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ίσα προγράμματα σε ό,τι αφορά τις άδειε τις γονεϊκές άδειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρουμε ότι όταν οι άντρες φροντίζουν τα παιδιά, θα είναι και πολύ πιο εμπλεκόμενοι στη ζωή των παιδιών και στη συνέχεια της ζωής τους. Και είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, το βλέπουμε, να έχουν μητέρε που δουλεύουν. Αν εδώ λοιπόν μιλάμε και για τις μελλοντικέ γενιές, και την καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού, ίσω είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τι επιχειρήσει το ζήτημα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε να δούμε και την... αυτό το βίντεο λέει η πρόεδρος.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 So just for information, system in the UK where the woman can give some of the leave to the man. Η ιδέα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα αφήνει μέρος της φροντίδας των παιδιών και στους άντρες, όπου η γυναίκα δεν είναι ο πρώτιστος. Και είναι ένας τρόπος όπου οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν προσαρμόζοντας λίγο τα δεδομένα, να ενθαρρύνουν τους άντρες να πάρουν μεγαλύτερη άδεια. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Βλέπω ότι υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Περνάμε τώρα στην Κάθριν Μίλλερ, πρόεδρος των, του Γυναικείου Συνδέσμου Δικηγόρων στην Ευρώπη. Very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Δύο Φύλων, ε, Κυρίες και κυρίες της ε, Γραμματείας, ε, διερμηνείς ε, και προσκεκλημένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σήμερα στην Ακροασία αυτή. Λέγομαι Κατερίνα Μίλλερ και είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Γυναικών Δικηγόρων. EULA. Είμαστε μη κυβερνητική ε, οργάνωση ε, κατοχωρισμένη στο Βέλγιο ως ε, μη κερδοσκοπική οργάνωση και είμαστε Ένωση Γυναικών Δικηγόρων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και των χώρων ΕΔΕΣ. Μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο. Σε όλο το κόσμο οι γυναίκες ε, αντιμετωπίζουν διάφορους, ε, ε, διάφορα εμπόδια στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, η λεγόμενη γυάλινη οροφή ή γυάλινη τύχη. Ε, χάνονται καθοδόν συχνά και γι' αυτό επικροτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το καυτό θέμα. ακούσαμε ότι είναι και πολύπλοκο θέμα. Κάτι που εξηγεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2017-2019. Από το 2017 και μετά, ο, Ευρω... ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για Ίση Αμοιβή προωθεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ίση αμοιβή. Πίσω, εκτός από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ε, κρύβεται και ο ΣΑ πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή που δείχνει πόσο ε, σοβαρά λαμβάνεται υπόψη παγκοσμίω ε, ο στόχο ίση αμοιβή μέχρι το 2030. Εξετάσαμε το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν ε, πολλές σημαντικές και κάποιες λιγότερο σημαντικές δράσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις βασικές πτυχές που πιστεύουμε ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι η ίση αμοιβή, όπως ανέφερε και η Vivian Hunt και οι άλλοι προλαλήσαντες, ε, είναι ένα business case. Σημαίνει ότι ε, θα έχει ωφέλη επιχειρηματικά. Οι στρατηγικές ε, ίσης αμοιβή ε, είναι σημαντικές σε μια επιχείρηση, αλλά είναι σημαντικό και για τους ε, καταναλωτές και αποτελεί σημαντικό τμήμα της μελλοντικής στρατηγικής επιχειρήσεων. Η Vivian Hunt αναφέρθηκε σε στοιχεία της McKinsey. Θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες κάνουν το 80% των καταναλωτικών αγορών, ελέγχουν πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και 29 τρισεκατομμύρια δολάρια προβλέπεται να περάσουν από τα χέρια τους τις επόμενες δεκαετίες. Οι γυναίκες έχουν οικονομικό σθένος και αγοράζουν προϊόντα που σέβονται τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης που συμπεριλαμβάνει και την ίση αμοιβή. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι το θέμα της κατανάλωσης είναι πολιτικό. Ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο εδώ. Πιστεύουμε ότι είναι να σπάσουμε τις παλιές δομές. Χρειαζόμαστε νέες δομές, καλύτερο σύστημα. Ε, το θέμα δεν είναι να επισκευάσουμε, να βελτιώσουμε τις γυναίκες. η είναι πολύ θετικό ότι βρίσκονται στην κορφή του θεματολογίου για την πολιτική και για τις επιχειρήσεις το θέμα το, της ισότητας. Αλλά ακόμα και οι γυναίκες που δεν ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία έχουν επιρροή, μπορεί, μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινωνία των πολιτών και μπορούν να καταναλώνουν συνειδητά κάθε απόφαση αγοράς είναι κάτι που έχει συνέπειες. Επίσης, η ίση αμοιβή είναι ένα θέμα νομικό. Επί της αρχής ήδη έχουμε αρκετούς διεθνείς και εθνικούς κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από όλους τους κύκλους ενδιαφερομένων ε, σχετικά με την ίση αμοιβή, ιδιαίτερα ε, το διάταγμα του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Υπαριθμών 100, που υιοθετήθηκε το 1951, που ε, υπογράφηκε από 173 κράτη. Όπως ανέφερε η Τίνα Άστολα, έχουμε και το κοινοτικό κεκτημένο. Όταν η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ το 1958, είχε μόνο μία διάταξη που ε, αφορούσε άμεσα την ισότητα των ε, δύο φύλων, την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών. Το άρθρο 119 είχε συμπεριληφθεί στη συνθήκη διότι η Γαλλία ήθελε να αποφύγει στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη-μέλη που ενδεχομένως να μην χρειάζεται να αμείβουν ίσα τις γυναίκες, κάτι που θα έδινε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στη Γαλλία. Ωστόσο, το 1956 το δικαστήριο ε, απεφάνθη ότι το άρθρο 119 είχε όχι μόνο οικονομικό στόχο, αλλά και κοινωνικό. Συνέβαλε στην κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Επαναλαμβάνω, ήδη το 1976 έγινε αυτό. Αργότερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο οικονομικός στόχος είναι δευτερεύον σε σχέση με τον κοινωνικό. Η ίση αμοιβή αποτελεί έκφανση ε, των μελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν γίνει πολλές νομοθετικές προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη μας. Μερικές είναι πιο φιλόδοξες, ε, άλλες λιγότερο. Ας εξετάσουμε την γαλλική νομοθεσία, όπου έχουν μεταφερθεί ήδη από το 1972 οι υποχρεώσεις για ίση αμοιβή στο Εθνικό Δίκαιο. Εννέα νόμοι έχουν υιοθετηθεί έκτοτε, ο πιο πρόσφατος το 2014, που μπορεί να θεωρηθεί πρότυπο. Ωστόσο, και στα 28 κράτη-μέλη, το μισθολογικό χάσμα συνεχίζει να υπάρχει με διακυμάνσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και παίρνω τώρα ε, στο τρίτο θέμα που θέλω να πω. Έχει να κάνει και με την ψηφιοποίηση. Ε, στις εποχές του γρήγορου μέλλοντος και της σκοτεινής πλευράς των δεδομένων ε, ε, είναι εύκολο να ε, ξεχάσουμε κάποιες ε, ομάδες. Για παράδειγμα, οι ε, μαύροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό αναγνώρισης προσώπων, διότι δεν αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους. Ή όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τις γυναίκες, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναγνωρίζουν μάλλον δεν αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκε ε, ε, δυσκολεύονται περισσότερο στη χρήση λογισμικού για την αναγνώριση φωνή από ότι οι άντρε, ε, διότι πολύ απλά το λογισμικό δεν αναγνωρίζει τόσο εύκολα τη φωνή του. Αυτό και πάλι οδηγεί σε χαμηλότερο ή καθόλου εισόδημα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την έρευνά του που υιοθετήθηκε το Ιανουάριο του 2017, περισσότερες γυναίκες κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της τεχνολογίας και οι γυναίκες αυτές έχουν λιγότερες ευκαιρίες να περάσουν σε θέσεις εργασίας υψηλότερων δεξιοτήτων, λέει η έκθεση. Ακόμα και με επανεκπαίδευση, οι γυναίκες έχουν λιγότερες επιλογές όσον αφορά ε, εναλλακτικές σταδιοδρομίες σε σχέση με τους άντρες. Περνώ τώρα στις συστάσεις μας. Ο σύλλογός μας ε, συστήνει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019. Εάν τα αποτελέσματα τη αξιολόγηση δεν είναι ικανοποιητικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνει εναρμονισμένη νομοθεσία για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα. Ανεξάρτητα, ο σύλλογό μα ε, θα επικροτούσε προσπάθειες από τα 28 κράτη-μέλη να ενισχύσουν ε, την νομοθεσία τους ε, και να αυξήσουν τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι επόμενες τρεις διατάξεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τέτοιες ε, νομοθετικές προσπάθειες. Πρώτον, είμαστε υπέρ του να κατονομάζονται οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται σε ιστοσελίδες των εθνικών κυβερνήσεων ή σε άλλες επίσημε ιστοσελίδες. Δεύτερον, προτείνουμε στην εθνική νομοθεσία να εισαχθεί δικαίωμα πρόσβασης σε ε, μισθολογικά στοιχεία δύο ανδρών τουλάχιστον και μια γυναίκα σε παρόμοια θέση για σύγκριση ε, των αποδοχών τους. Επίσης, ε, θα επικροτούσαμε τη δυνατότητα ε, συλλογικών αγωγών, κάτι που θα βελτιώσει τις δυνατότητες ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσφύγουν σε περιπτώσεις μη ίσης αμοιβή. Επίσης, θα ήθελα τώρα να περάσω στο σχέδιο δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσιάσει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων του Progress. Ε, θα θέλαμε να συμπεριληφθεί και πρόγραμμα ε, του 2014-2016 που δημιουργήθηκε για να ε, προωθηθούν οι δυνατότητες των γυναικών. Στο πρόγραμμα αυτό θα βρείτε όλες μας, όλες μας τις συστάσεις. Επίσης, η Ιούλα, η οργάνωσή μας, θα ήθελα να σας συγχαρεί για την κοινή προσπάθεια ε, για την πραγματοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Δυστυχώς όμως πρέπει να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας ε, σχετικά με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου ε, πάνω στην οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, διότι πιστεύουμε ότι έχει αποδυναμωθεί η νομοθεσία. Ε, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσουν, ωστόσο με, λιγότερο, με χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας από ό,τι πριν. Εναπόκειται λοιπόν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασώσει ε, την φιλόδοξη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου 2017. Ε, ε, δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη οι στόχοι. Ε, η οργάνωσή μα, η Γιούλα, είναι διατεθειμένη να σα στηρίξει στη διαδικασία αυτή. Και κλείνω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ βιωσιμότητα χωρίς ίσες αποδοχές, χωρίς ισότητα. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να ε, δημιουργήσουμε ένα μέλλον για την ανθρωπότητα ε, σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιο θέλουμε να είναι το μέλλον μας. Εάν μπορούσαμε να Εφόσον μπορέσαμε να εφαρμόσουμε την ε, οδηγία για την προστασία των δεδομένων με τόση αντίθεση που υπήρχε, θα πρέπει να μπορούμε να πετύχουμε και ίση αμοιβή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα εμψυχωτικά σας λόγια και την υποστήριξη που δώσατε στο πακέτο μέτρων για, την, για το συνδυασμό προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Μάλιστα. Επανερχόμαστε τώρα στη συζήτηση με την Ομιγύρη. Έχετε την ευκαιρία τώρα να θέσετε τις ερωτήσεις ε, στις καλεσμένες από τα πάνελ. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. κυρία Κριστίνα Μορβάη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες ε, των καλεσμένων μας. Ε, δεν ακούω όμω ε, ουγγρική διερμηνία. Υπάρχει δυνατότητα. Θα ήθελα, θα προτιμούσα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Α, ωραία. Υπάρχουν και ουγγρικά a, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω την εξής ερώτηση. Από τους ε, σημερινούς εμπειρογνώμονες αναφέρθηκε το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών και τονίστηκε ότι υπάρχει σημαντική διάκριση εις βάρος των γυναικών. Θα ήταν δυνατόν κάποια από εσά να μας πει, για παράδειγμα η κυρία από το Δικηγορικό Σύλλογο, να μας πει πώς έχει η κατάσταση στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Πολύ σωστά αναφέρθηκε η πρόταση για τον, το να κατονομάζονται οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται, να δημοσιεύονται τα ονόματα των επιχειρήσεων που κάνουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στο μισθολογικό τομέα. Μήπως θα ήταν δυνατόν να δημοσιεύουμε και ονόματα επιχειρήσεων στα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη ή στα πιο φτωχά που κάνουν τις διακρίσεις αυτές. Διότι εδώ η διάκριση βάρους των γυναικών είναι διπλή. Γνωρίζετε ότι μία πολίτρια εντός της ίδιας επιχείρησης στη δική μου χώρα λαμβάνει πολύ χαμηλότερο μισθό από ότι οι συναδέλφισές της στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση και αυτή είναι μια αρνητική διάκριση. Επιπλέον θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι Όταν επιδεικνύουμε αλληλεγγύη όπως εδώ, διαπιστώνουμε ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν ε, την κατάσταση ότι τα παιδιά τους εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Προσελκύουν τους νέους ε, τα κράτη-μέλη που μπορούν να προσφέρουν ε, καλύτερες αμοιβέ και συνθήκες. Ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, κατά τις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πολλοί νέοι εγκαταλείπουν ε, τις χώρες τους για να πάνε στις πλουσιότερες χώρες. Αλλά είναι και θέμα φτώχειας, διότι οι γυναίκες των οποίων τα παιδιά εγκαταλείπουν τη χώρα τους τελικά μένουν πίσω με πολύ χειρότερες οικονομικές συνθήκες. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω όσον αφορά την Ουγγαρία και την Πολωνία. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση για πολιτικούς λόγους. Βλέπουμε ότι κάποια κονδύλια αφαιρούνται από τις χώρες αυτές και έτσι οι διαφορές Ανατολής και Δύσης ε, γίνονται πιο οξύες. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχουν να πούνε σχετικά με τα θέματα αυτά οι ομιλητριέ μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανεί άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, μια και έχω και πολωνική διερμηνία, θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιε ερωτήσει, αλλά θα τι κάνω στη μητρική μου γλώσσα. Καταρχήν, να ξεκινήσω με ευχαριστίες. Ευχαριστίες προς τις εμπειρογνώμονες που με έδωσαν το παρόν στη συζήτηση, γιατί ήταν πολύ συναρπαστική συζήτηση, πηγή έμπνευση ε, και πολύ ελπιδοφόρα αυτά που ακούσαμε για πολλά παραδείγματα που στέφθηκαν με επιτυχία και πολλές δράσεις που σημείωσαν πραγματική πρόοδο. Καταλάβαμε ότι είναι δυνατή η πρόοδος. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικώ στις πολιτικές ομάδες ε, δεν ε, βλέπουμε πάντα απτή πρόοδο, γιατί δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των διατάξεων που θεσπίζουμε σε νομοθετικό επίπεδο. Χαίρομαι όμως που βλέπουμε εδώ κάποιες ε, απτές ε, ε, εξελίξεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τις εκπροσώπους ενώσεων ή επιχειρήσεων. Έχετε απτές αποδείξεις ότι οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που επέλεξαν οι εταιρείε είναι αποτελεσματικές. Έχετε επίσης εταίρους στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, γιατί οι επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε έχουν έδρες ε, και παραρτήματα σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε συνεργάζεστε επί τόπου με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ή οι δρασει σας περιορίζονται στις ε, μεγάλες πολυεθνικές ε, και είναι μόνο μεμονωμένες οι περιπτώσεις αυτές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, πριν από μερικά χρόνια οργανώσαμε στην Πολωνία με εμπειρογνώμονε τη αγορά εργασία. αντίστοιχη δημόσια κρόαση και ακούσαμε τότε από εμπειρογνωμονε, άνδρες και κυρίω γυναίκε ότι για, για πολλά χρόνια 15-20 ε, χρόνια ανάλυσης ε, του μισθολογικού χάσματος ε, διαπίστωσαν ότι ακριβώς αυτές οι μισθολογικές διακρίσεις ήταν από τα πιο σοβαρά προβλήματα που οφείλονταν στην νοοτροπία την εταιρική η εταιρική κουλτούρα μπορεί να μην είναι κάτι ορατό από τους πολιτικούς, αλλά η κουλτούρα είναι υπεύθυνη για αυτές τις ανισότητες και για αυτές τις μυθολογικές και άλλες διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα στις ε, εταιρείε. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί αυτό το θέμα της ε, επιχειρηματικής, της εταιρική νοοτροπίας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι δυσπρόσιτη αυτή η έννοια της νοοτροπίας. Γι' αυτό θα πρέπει με νομοθετικό τρόπο να εφοδιάσουμε τις εταιρείες με μηχανισμούς που να τους επιτρέψουν να αλλάξουν αυτή την κουλτούρα που επικρατεί στις σε αυτή την οτροπία. Μερικές το κατάφεραν, όπως εσείς, οι ε, δικοί σας, η Υπάρχουν και άλλες που εφάρμοσαν αντίστοιχες διαδικασίες ή είστε μόνο εσείς κάποιες ε, νησίδες, κάποιες οάσεις πρόοδου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις, ε, των γυναικών που είπατε ότι πολλές φορές θα πρέπει να σταματήσουμε να λάβουμε απόσταση και να επικεντρωθούμε στις γυναίκες κυρίως. Και επίσης ε, να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις γυναίκες κρατώντας ε, τα χαρακτηριστικά τους να επιτύχουν την προσωπική τους και την επαγγελματική τους ε, αυτοεκπλήρωση. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω τώρα το λόγο στις καλεσμένες μας ε, και από το δεύτερο πάνελ πρώτο και μετά από το πρώτο για να απαντήσω σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Καταρχήν να απαντήσω στην πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όταν εξετάζουμε τι μισθολογικέ διακρίσει, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποιε γυναίκε είναι σε πολύ ε, μειονεκτική θέση, είτε λόγω τη εθνότητά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε λόγω τη επικότητά του, είτε λόγω τη ηλικία του. Και σίγουρα οι μισθολογικέ διακρίσει είναι μεγαλύτερη βάρο των γυναικών. Αλλά και γυναίκε, ιδιαίτερα κάποιων μειονοτήτων, εθνοτικών ή άλλων, αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερε διακρίσει και προκλήσει. Και οι πολιτικές είναι κλειδί, αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Σίγουρα δεν υπάρχουν α, α, κρατικές πολιτικές, θα πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ, αλλά χωρίς αλλαγή νοοτροπίας δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αυτές οι ε, πολιτικές. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την έρευνά μας, να δούμε τι πρακτικές θα επιφέρουν τη διαφορά. Και το θέμα της κουλτούρας, της νοοτροπίας είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και η Έμα. Ε, θα Σίγουρα οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερες ε, υποχρεώσεις και δεν μπορούν να καθίσουν στο σπίτι μέχρι αργά όπως κάνουν οι άντρες. Έχουν ε, να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν όλη αυτή την κουλτούρα να την αλλάξουμε και φυσικά οι διευθύνοντες σύμβουλοι να στενιστούν αυτές τις νέες πολιτικές και να δώσουν το καλό παράδειγμα, να γίνουν υποδείγματα. Επίσης, οι εταιρείε θα πρέπει να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις. Και στο Business in the Community, στη δική μας οργάνωση, έχουμε καταπληκτικούς εργοδότες που μας έχουν δείξει ε, τι μηχανισμός ε, ε, λειτουργεί. Για παράδειγμα, έχουμε εταιρείε που έχουν δώσει ίσες ευκαιρίες γονικής, άμυνα, γονικής άδειας με τις ίδιες αποδοχές σε άνδρες και γυναίκες και έχει αυξηθεί κατά 12% η λήψη τέτοιων γονικών αδειών και από τους άνδρες. Τέτοιες πρακτικές τις προσπαθούμε να τις διαδώσουμε και σε άλλες εταιρείε, αλλά και στις κυβερνήσεις για να λάβουν αντίστοιχε δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ σε μερικά από τα σχόλιά σας και να προσυπογράψω αυτά που είπε η Κλώε. Φυσικά, εγώ εκπροσωπώ εδώ έναν εργοδότη, εργοδότη από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, και θεωρώ ότι οι εργοδότες έχουν μείζωνα ρόλο να διαδραματίσουν. Εγώ αφιέρωσα πολύ χρόνο στη συζήτηση με άλλε εταιρείε, εξηγώντα τι έχουμε κάνει εμεί στην Deloitte, ε, και μάλιστα έχουμε δημιουργήσει πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών και στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες με πολύ ανοιχτό τρόπο σε όποιον ενδιαφέρεται και παρουσιάζουμε τις, ε, τα επιτεύγματά μας και το θεωρώ αυτό θέμα των ευθυνών μου, των καθηκόντων μου. Επίσης, το θέμα της ε, διαδικασίας. Ε, έχουμε τις παραδόσεις των εταιριών και την οτροπία και την κουλτούρα. Συμφωνώ και το είπα και προηγουμένως στην ομιλία μου, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το χώρο εργασίας. Και μέσα στα χρόνια της λειτουργία μας έχουμε δημιουργήσει πολλά πολλές πρωτοβουλίες όπως ε, πάνελ πρόθεσης για να δούμε αν κάποιος είναι έτοιμος και γι' αυτό έχουμε πάνελ, αλλά τα περισσότερα πάνελ ήταν ανδροκρατούμενα. Ε, έχουμε λοιπόν άλλες διαδικασίες που διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργούσαν. Ε, δεν ήταν αρκετά περιεκτικές γιατί απέκλειαν κάποιες μειονότητες. Επίση, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρηματίσει. Σίγουρα ο ρόλο των επιχειρήσεων φτάνει μέχρι τα σχολεία για να αποφευθεί ο διαχωρισμό που υπάρχει και που φαίνεται στην έκθεση και στι συστάσει. Μάλιστα, το 2016 κάναμε μια σχετική έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάσαμε ποιε είναι οι ρίζε του μισθολογικού χάσματο. Ήταν πραγματικά συναρπαστική η έρευνά μα και έδειξε με σαφήνεια ότι οι ρίζε ε, των μισθολογικών διακρίσεων ε, βρίσκονται στι επιλογέ που κάνουν τα κορίτσια στο σχολείο. Και το λέω μητέρα 9 χρονών διδήμων, που βλέπω ήδη να προδιαγράφονται κάποιε επιλογέ και βλέπω ήδη κάποια στερεότυπα. Σε κάθε στάδιο υπάρχει μια επιλογή που θα πρέπει να γίνει ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, από το σχολείο μετά στο πανεπιστήμιο και τα κορίτσια οι γυναίκες επι, επιλέγουν να απομακρυνθούν από τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τους υπολογιστές. Γιατί είδαμε πόσο, σημαντικές θα είναι, σημαντικοί θα είναι οι υπολογιστές στι μελλοντικέ θέσει εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε και τα κορίτσια προ τέτοιου είδου σπουδέ. Αλλιώ, θα συνεχίσουν να κάνουν επιλογέ μακριά από τι θετικέ επιστήμες και οι εταιρείε θα μπορούσαν με εταιρικέ σχέσει να βοηθήσουν για να διαμορφώσουν κάποια ε, ιδεώδη, κάποια ε, υποδείγματα, ε, κάποια πρότυπα για να αλλάξουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό των κοριτσιών. Οπότε, εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη και οι εταιρείε να συνεργαστούμε με τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και με την κυβέρνηση για να αλλάξουν αυτά τα στερεότυπα και αυτή η νοοτροπία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καταρίνα Μίλλαρ και πάλι. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ μια μη κυβερνητική οργάνωση. Οπότε η απάντησή μου θα είναι κάπως διαφορετική. Δεν εκπροσωπώ εταιρεία ή επιχείρηση. Ε, ήμουν το Μάρτιο στην Επιτροπή της Νέας Υόρκης για την κατάσταση των γυναικών και συμμετείχα στην αντιπροσωπεία της γερμανικής κυβέρνησης και συμμετείχα σε μια συνάντηση για την ε, ισότιμη αμοιβή. Και όλες, όλα τα μέλη της στη συνάντηση είπαν δεν ξέρουμε τι λειτουργεί. Δεν το ξέρουμε γιατί πραγματικά δεν λειτουργεί. Εσείς είπατε ότι κάτι συμβαίνει με τα παιδιά μας ήδη από την πολύ μικρή ηλικία, από την ε, παιδική ηλικία. Όταν ρωτάμε τα παιδιά 4 χρονών ε, τα κορίτσια, τα γόρια και τους λέμε τι θέλουν να γίνουν, θέλουν να γίνουν ε, ήρωες, Superman, Superwoman. Μετά από μερικά χρόνια τα γόρια εξακολουθούν να δίνουν την ίδια απάντηση, ότι θέλουν να γίνουν ε, ήρωες, Superman. Ενώ οι γυναίκες, τα κορίτσια αρχίζουν και στρέφονται προς άλλες ε, κατευθύνσεις. Θέλουν να αναλάβουν τη φροντίδα, να γίνουν μοντέλα, να γίνουν μητέρες. Κάτι αλλάζει λοιπόν στην, στον προσανατολισμό τους των επαγγελματικών και είναι δύσκολο να αλλάξει η κουλτούρα μιας εταιρεία, η νοοτροπία μιας εταιρεία. Είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται πραγματικά η έντιμη δέσμευση των διευθυντών και του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση του, των ηγετικών στελεχών, δεν πρόκειται να έχουμε μία ορατή λύση, μια πρόοδο. Μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω να λειτουργεί τίποτα άλλο. Και ευχαριστώ για την ερώτηση, ναι, το έχουμε υπόψη μας. Ήταν πολύ περίπλοκη, πολύ σύνθετη μάλλον η ερώτησή σας και παρόλο που είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας δώσω εκτενή απάντηση. Εγώ σας παραπέμπω στο κράτος δικαίου. Από τη στιγμή που έχουμε μια νομοθεσία στην Ουγγαρία που προβλέπει ότι μπορούμε να κατονομάσουμε τις επιχειρήσεις, να τις δακτυλοδείξουμε, τότε γίνεται. Αν δεν είναι νομότυπο κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο. Οπότε εξαρτάται από το νομοθέτη, από την εθνική νομοθεσία, από την εθνική νομιτάξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο. Ε, στην Ευρώπη η οργάνωσή μας συνεργάζεται με, τη, με το ουγγρικό μας μέλος και διαπιστώνουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, στην Ουγγαρία είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί μερικές φορές οι ουγγρικές εταιρείε ε, μπορεί να δημοσιεύουν τα στοιχεία τους, αλλά κανένας ε, δεν ενδιαφέρεται. Η εταιρεία είναι κλειστή, υπάρχουν στεγανά. Και για την Ουγγαρία είναι πολύ σημαντικό ε, να έχουμε στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, το ίδιο έκανε και στην Ισπανία και στη Βουλγαρία. Και είδα ότι για τι χώρε αυτέ είναι πολύ σημαντική η εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και καλό θα ήταν να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε από κοινό όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τίνα Άστολα, που είναι Γενική Διευθύντρια τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο εξετάσαμε την κατάσταση συγκριτικά μεταξύ των νέων και των παλαιών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα ότι το παράδειγμα δείχνει ξεκάθαρα πόσο τα δεδομένα αλλάζουν τα, τα δύο φύλλα. Επομένως, σε κάθε δουλειά που ξεκινάμε να κάνουμε, θα πρέπει να κοιτάμε τις επιπτώσεις που έχει η νομοθεσία στις γυναίκες. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι το κάνουμε αυτό. Παράλληλα, πιστεύω ότι σε αυτό το σχέδιο δράσης που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, δηλαδή δεν υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες ε, μεταξύ των διαφορετικών χωρών, σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με τις οικονομικές διαφορές και στα διάφορα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτιστικό, το ζήτημα κουλτούρας, θα συμφωνήσω με όλους όσους μίλησαν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τα παιδιά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ε, σε διάφορες εταιρείες στον δημόσιο τομέα. Ακούσαμε και την ομιλία από τον Deloitte. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν από πάνω όμως οι αλλαγές. Και από, όλους, από όλα τα άτομα που βρίσκονται σε ηγετικέ θέσει, νομίζω ότι είναι σαφέ ότι μιλάμε σοβαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, κυρία Διευθύντρια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Vivian Hunt από την εταιρεία McKinsey. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Χάντ. Ένα κοινό σημείο μεταξύ των διαφόρων ερωτημάτων σε σχέση με τη νομική θέση των επιχειρήσεων και τις κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και στα διάφορα παραδείγματα και πόσο πολύ ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να επηρεαστεί, είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη από πραγματικά δεδομένα, στοιχεία. Αυτό ισχύει και όταν χαράζει κανείς πολιτική και αυτό ισχύει και για τις εταιρείε και για τους υπαλλήλου τους. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε και να κινηθούμε προς εκθέσεις και αναφορές που βασίζονται σε δεδομένα σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και τις αμοιβέ τους. Βεβαίως και είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε τη δική μας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει και όλες τις, όλα τα κρατημέλη που, είναι, που απαρτίζουν την οργάνωσή μας. Από μαζί με την Επιτροπή για τις Γυναίκες και την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και την Επιτροπή για την Οικονομική Παραγωγικότητα. Να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα για να μπορέσουμε να βρούμε την λύση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα στην Ιταλία, στην Ουγγαρία κτλ. Διότι βεβαίως δεν υπάρχει ένα μέτρο που να μπορεί να λειτουργήσει παντού. Το δεύτερο σημείο που χρειαζόμαστε απτά δεδομένα έχει να κάνει με τις πολιτικές και τις πρακτικές. Μόνο αν μπορέσουμε να εξετάσουμε κάποια πράγματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μόνο τότε θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τα 4-5 πράγματα που κάθε είτε τομέας του δημοσίου είτε εργοδότης πρέπει να κάνει. Και είναι ανάγκη να έχουμε στοιχεία από τις ίδιες τις εταιρείες για να μπορέσουμε να διακρίνουμε ποιες είναι αυτές οι μία, 2, 3, 4 δράσεις που θα έχουν τι, το, το, πιο αποτελεσματικό, τις πιο αποτελεσματικές επιπτώσεις. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα λίγα πράγματα που θα μπορούν να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα να αποφασίσουμε ποιε θα είναι οι επιχειρησιακές παρεμβάσει, ή οι παρεμβάσει σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και πάλι όμως έχουμε ανάγκη από αυτά δεδομένα για να δούμε πού μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα. Το τρίτο σημείο που είναι ανάγκη να κλείσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ ανεκδότων και απτών στοιχείων από τη δική μας εμπειρία στη Μακέντζη μπορώ να σας πω ότι κάθε ε, περίπτωση που έχουμε εξετάσει που ήταν ποσοτική και αφορούσε 15 εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούσε να προσεγγίσει συστηματικά το ζήτημα της κουλτούρας. Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, 80% των περιπτώσεων έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κουλτούρα του εργοδότη και όχι του εργαζομένου. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που καταφέρνουμε να κλείσουμε αυτό το χάσμα στην κουλτούρα αν έχουμε το κουράγιο να κοιτάξουμε τα δεδομένα ως έχουν. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω, όπου και πάλι θεωρώ ότι χρειαζόμαστε από τα δεδομένα, έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Πολλές εταιρείε, πολλοί από αυτούς που χαράζουν πολιτική προσπαθούν να κάνουν ένα πράγμα ωστόσο καταλήγουν να πνίγονται από, τα, από, τους, από τις παραμέτρους και να μην έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Πολλές από τις εταιρείε όμως που έχουν θετικά αποτελέσματα, αυτό που πρέπει να κάνουμε, να, να συγχαίρουμε τις εταιρείε που έχουν διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ, να θέτουν το καλό παράδειγμα. Μια βάση δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τη ε, συστηματική εξέταση, ενθάρρυνση των εταιριών που τα πάνε καλά σε αυτό το τομέα, πιστεύουμε θα συμβάλλουν τα μάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ingrid τώρα από το Αυστριακό Επιμελητήριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με το μισθολογικό χάσμα. Καταρχάς βλέπουμε και εμείς από τις στατιστικές ότι οι γυναίκες μετανάστες βγάζουν λιγότερα από τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί στην Αυστρία. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το χάσμα. Έτσι, αλλά επίσης στην Αυστρία αλλά και σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι ότι χρησιμοποιείται φτηνό εργατικό δυναμικό. για παράδειγμα στην φροντίδα ηλικιωμένων 24 ώρες το 24ωρο. Βλέπουμε ότι εργάζονται γυναίκες από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Και οι γυναίκες αυτές εργάζονται με χειρότερες συνθήκες εργασίες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μισθολογική πίεση. Άλλο θέμα είναι η κουλτούρα στις επιχειρήσεις, η νοοτροπία. Ακούσαμε το θέμα των ε, μισθολογικών εκθέσεων και της διαφάνειας. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο το θέμα αυτό, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αμοιβή ανδρών και γυναικών. Όταν υπάρχει πλήρης διαφάνεια, γίνεται αξιολόγηση και της εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διάφορες δραστηριότητες αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. Και υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να ε, οδηγήσουν αυτές οι εκθέσεις σε τριβές εντός της επιχείρησης. Όσον αφορά λοιπόν ε, την κουλτούρα εντός των επιχειρήσεων, όσο έχουμε μόνο κάποιες λίγες γυναίκες σε έναν ανδρικό κύκλο είναι πολύ δύσκολο να αισθάνονται άνετα. Πολλές γυναίκες μπορεί να βρεθούν σε διευθυντική θέση ή να έχουν τεχνική εκπαίδευση, εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες, αλλά τελικά να εγκαταλείψουν τις θέσεις αυτές επειδή δεν νιώθουν πολύ άνετα. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Γιατί μας πιέζεται τόσο με το χρόνο αφού είμαστε μόνο δύο ευρωβουλευτές. Θέλω μια διευκρίνηση. Εγώ δεν μιλώ για τις μετανάστριες. Μιλώ για τις γυναίκες που είναι Ευρωπαίοι πήκοοι, έχουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και η κανονικά πρέπει να είναι ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες με τους Αυστριακούς, με τις Αυστριακές και παρόλα αυτά κερδίζουν τρεις φορές λιγότερα χρήματα για την ίδια θέση και μάλιστα απασχολούνται από την ίδια εταιρεία που πολύ συχνά είναι Αυστριακή εταιρεία. Μακάρι θα ήταν, ε, θα ήταν ευχής έργο ε, να είχε διορθωθεί αυτή η κατάσταση τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί το 2004 μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να νιώθουμε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. ακόμη και οι μετανάστριες που πηγαίνουν στην Αυστρία για να δουλέψουν δεν είναι μετανάστριες από τον τρίτο κόσμο. Είναι από την Ουγγαρία, από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έπρεπε να κερδίσουν το ίδιο με τους Αυστριακούς, με τις Αυστριακές. Και καλό θα ήταν αυτή την αλληλεγγύη που νιώθετε για τι άλλε γυναίκε να την νιώθετε και σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δυστυχώ πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δημόσια ακρόασή μα. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμότατα τι καλεσμένε μα, εμπειρογνώμονε που μα παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσε θέσει. Μα έδωσαν πραγματικά έμπνευση με τα σχόλιά τους για την εξάλληψη των μισθολογικών διακρίσεων το πιο σημαντικό που ανέκυψε από την ακρόαση είναι η δυνατότητα να κατανικήσουμε αυτό το μισθολογικό χάσμα, γιατί πραγματικά πριν από την ακρόαση ήμουν κάπως απεσιόδοξη. Τώρα ε, έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι εφικτή η κατάρρευση των μισθολογικών διακρίσεων και η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος. Απλώς χρειάζεται να συμπληρώσουμε τις δυνάμεις μα, Οι επιχειρήσει, οι κυβερνήσεις και όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε από κοινού να καταπολεμήσουμε αυτό το κενό. Και σίγουρα οι νομοθέτες θα διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο σε αυτό το θέμα αλλά και η επιχειρηματική, οικονομική διάσταση και προοπτική ίσως διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάλληψη των μισθολογικών διακρίσεων, γιατί το επιχείρημα της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό και βάσιμο. Αλλά ε, μερικές φορές το αντεπιχείρημα είναι το οικονομικό αυτό επικαλούνται μερικοί. Χαίρομαι που ούτε το οικονομικό επιχείρημα δεν συμβάλλει υπέρ της διαιώνισης του μισθολογικού χάσματος. Ίσα ίσα το αντίθετο. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση, αλλά και βούληση αλλαγή σε επίπεδο επιχείρησης. Και χωρίς αυτή τη βούληση, την επιθυμία αλλαγή, δεν πρόκειται να έχουμε αλλαγή τη κατάσταση. Και σίγουρα ο, σημαντικός, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η επιχειρηματική εταιρική κουλτούρα, η εταιρική νοοτροπία και αυτό προϋποθέτει μια επιθυμία αλλαγής, μια βούληση αλλαγής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλαγή και στη διαχείριση και στη ηγεσία, στη διεύθυνση. Θα πρέπει τα ηγετικά στελέχη τη επιχείρηση ε, να είναι ευαισθητοποιημένα στην ανάγκη τη υλοποίηση ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και σε μισθολογικά θέματα. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά θα είμαστε πολύ κοντά στην επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν του τους συμμετέχοντες, τις συμμετέχους μάλλον στην δημόσια κρόση και ολοκληρώνουμε αυτό το τμήμα της συνεδρίασης. Yeah.

Okay. Um, Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ακούσουμε την πρέσβυρα της Ισλανδίας, ε, μιας χώρας που είναι, έχει τα πρωτεία παγκοσμίω ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Θα ακούσουμε την κυρία Μπέρντις Έλερστότηρ που θα μας κάνει την εισαγωγική ομιλία. Εγώ, η κυρία Χέντ, είμαι αντιπρόεδρος της ΣΥΝΕΑ, της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την ε, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Θα μας πει η πρέσβη της Ιρλανδίας ε, τα περισσότερα στην Ισλανδία και γιατί οι συντονιστές αποφάσισαν να εκπροσωπήσουν τις ε, χώρες αντιπροσωπείας η νέα, δηλαδή Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε μια ανταλλαγή απόψεων για να μας παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σε θέματα ισότητας φύλων. Και αυτό θα δώσω το λόγο, όπως είπα, πρώτο στην πρέσβυρα της Ισλανδίας, την κυρία Έλερ Έλερστότυρ, για να μας πει πώς τα κατάφερε η Ισλανδία και έχει τόσο καλές επιδόσεις στην ισότητα των φίλων; Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ε, είναι χαρά μου, όπως πάντα, να βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό βήμα για μας. Ε, δεν ε, βρισκόμαστε εδώ πολύ συχνά. Είναι λοιπόν τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας. Καταρχάς, θα μιλήσω λίγο για την ε, νέα νομοθεσία για την ίση αμοιβή αντρών και γυναικών και από ό,τι κατάλαβα μόλις είχατε σχετική ακρόαση. Μπορεί λοιπόν να σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην αύξηση του αριθμού και της επιρροής των γυναικών στην πολιτική και το δημόσιο βίο. Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, βία εις βάρος των γυναικών και να σας εξηγήσω πώς θέλουμε να πετύχουμε τη συμμετοχή των ανδρών στον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων και τέλος να αναφερθώ και στις σχέσεις Ισλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας ε, ένα σημαντικό γεγονός στην Ισλανδία που ήταν ε, κεντρικό στην ιστορία μας όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων που ήταν η απεργία των γυναικών στις 24 Οκτωβρίου του 1975. Χιλιάδες γυναίκες, το 90% του γυναικείου εργατικού δυναμικού εγκατέλειψαν την εργασία τους, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να απαιτήσουν περισσότερη ισότητα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι τότε η αμοιβή του αντιστοιχούσε στο 60% των γυναικών και υπήρχαν μόνο τρει γυναίκε βουλευτέ τότε. Είναι απίστευτο το ότι αυτό συνέβη τόσο πρόσφατα. Η ημέρα αυτή της γυναικείας κινητοποίησης ήταν επιτυχία, διότι αυτή η κινητοποίηση παρέλυσε την κοινωνία για μία μέρα, κάτι που έδειξε ότι η συμβολή των γυναικών στην οικονομία και την κοινωνία δεν είναι λιγότερο σημαντική από αυτή των ανδρών. Όπως είπα λοιπόν, ε, ήταν κεντρική στιγμή στην ιστορία μας η κρίσιμη μάζα γυναικών που συμμετείχε. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα και οι ομιλίες που έγιναν φάνηκε να ενδυναμώνουν σημαντικά τις γυναίκες στον αγώνα τους. Ε, όπως όμως και τόσα άλλα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την ιστορία δεν ε, συνέβη σε κενό αέρος. Ε, είχε να κάνει με εξελίξεις που συνέβησαν και πριν και μετά. Έχει βελτιωθεί από το 1975 η κατάσταση όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα. Ωστόσο δεν έχει εξαφανιστεί το μισθολογικό χάσμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν στοχευμένες δράσεις για να το εξαλείψουμε και να διατηρήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Τι πρόοδος όμως έχει σημειωθεί και τι δράσεις αναλαμβάνουμε. Ανάλυση του μισθολογικού χάσματος στην ε, Ισλανδία δείχνει ότι το χάσμα μειώνεται στο διάστημα 2008 έως 2016 το 2008 ερχόταν σε 6,6% ενώ είχε μειωθεί σε 4,5% το 2016. Ε, έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος, βλέπουμε όμως ότι είναι και επίμονο το μισθολογικό χάσμα εις βάρος των γυναικών. Και ε, βλέπουμε περισσότερους άντρες σε ηγετικές θέσεις όπως και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να έχουν ε, θέσεις μερικής απασχόλησης και να κάνουν περισσότερη μη ε, αμοιβόμενη δουλειά ε, στην φροντίδα άλλων ατόμων και στην κοινωνία. Βλέπουμε ανισορροπίες όσον αφορά τις δυνατότητες σταδιοδρομικής εξέλιξης και όσον αφορά τις συντάξεις η συμβολή των γυναικών είναι στα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι χαμηλότερη από ό,τι είναι των ε, ανδρών λόγω των ανισορροπιών. Η ομάδα εργασίας ε, για το μισθολογικό χάσμα συστήθηκε με διάφορους στόχους, ένας εκ των οποίων ήταν να παρακολουθούν την εφαρμογή πιλωτικού προγράμματος ε, για ένα Ισλαδικό πρότυπο ίσης αμοιβή. Και εν συντομία, Πρόκειται για ένα πείραμα για προώθηση ε, πειράματος ε, και από την 1η Ιανουαρίου φέτος το πρότυπο ίσης αμοιβή αποτελεί νομοθετική υποχρέωση με την οποία επιχειρήσεις ε, και άλλοι οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 25 άτομα πρέπει να ε, έχουν επιστοποίηση του, συστήματος, ε, του μισθολογικού του συστήματος. Στόχος είναι να αναπτυχθούν τα μισθολογικά συστήματα σύμφωνα με τις αρχές ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Η πιστοποίηση των συστημάτων αυτών προβλέπεται σε ένα διάστημα τριών ετών και στόχο έχει να πληρεί τις ε, απαιτήσει για ίση αμοιβή και στην νομοθεσία μας, ε, αλλά και στη, σε διεθνή όργανα, όπως είναι η Σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Νομοθεσία δεκαετιών ε, απαγορεύει τις διακρίσεις θα πρέπει να εφαρμοστεί όμως. Καταλαβαίνετε ότι έχει συζητηθεί πολύ το θέμα αυτό στην Ισλανδία. Τελικά όμως οι περισσότεροι βουλευτές συμφώνησαν ότι οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Η νέα αυτή νομοθεσία λοιπόν κάνει την Ισλανδία την πρώτη χώρα στον κόσμο που απαιτεί η πιστοποίηση του μισθολογικού συστήματος με βάση ένα υποχρεωτικό πρότυπο. Και έτσι η ε, ευθύνη μεταφέρεται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη. Πολύ ήθελα να ήμουν εδώ κατά την ε, συζήτησή σας. Ε, δεν ε, μπόρεσα να είμαι εδώ κατά τη συζήτησή σας. Αν έχετε ερωτήσεις όμως, πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω. θα ήθελα να αναφερθώ και στη θέση των γυναικών στην πολιτική και στο δημόσιο βίο. Κάποιοι από σας μπορεί να γνωρίζουν ότι η Κατρίν Ιάκοψ τότε είναι αρχηγός της κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία μας μετά από τις κοινοβουλευτικές τον Οκτώβριο του 2016 είδαμε πολύ σημαντική αύξηση της εκπροσώπησης γυναικών στο Κοινοβούλιο από 40 σε 48%. Επιτέλους λοιπόν 100 ε, ε, χρόνια μετά την έρξη των αγώνα των γυναικών μιλάμε για ισότητα στην πολιτική. Ένα χρόνο μετά όμως, τον Οκτώβριο του 2017, είχαμε προώρες εκλογές και μειώθηκε το ποσοστό. Οι γυναίκες λοιπόν τώρα αποτελούν το 38% των βουλευτών. Ε, είναι λοιπόν ένας συνεχής αγώνας. Ιστορικά η προώθηση της εκπροσώπησης των γυναικών οφείλεται στις ε, ε, ακούραστες προσπάθειες του κινήματος των γυναικών και τις προσπάθειες ε, γυναικείων ε, κομμάτων. Τη δεκαετία του 80 ήταν ε, πολύ χαμηλή η εκπροσώπηση των γυναικών. Μέχρι τότε το 2 έως 5% των βουλευτών ήταν γυναίκες. Το 1908 η πρώτη γυναίκα εξελέγει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ το 1922 εξελέγει στο κοινοβούλιο μας. Αυτό το πολιτικό πείραμα ε, ε, ε, επαναλήφθηκε το 1980, όπου είδαμε πάλι ραγδαία αύξηση των γυναικών. στην αγορά εργασίας της Ισλανδίας υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών, 80%. Ε, Ωστόσο, η εκπροσώπησή τους σε υψηλές θέσεις εργασίας και στο κοινοβούλιο είναι χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Επίσης βλέπουμε ότι ε, οι τομείς ε, όπου δεσπόζουν οι γυναίκες γενικά αμείβονται χαμηλότερα από ότι οι ανδρικοί τομείς. Επίσης έγιναν προσπάθειες να τροποποιηθεί ε, το επιχειρηματικό δίκαιο στην Ισλανδία ε, και να διασφαλίζεται το, ότι το 40% των μελών ε, των διοικητικών συμβουλίων αποτελείται από γυναίκες. Αυτό λοιπόν υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο το 2013. αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για δημόσιους φορείς πριν από αυτό. Οι γυναίκες ε, δεν ήταν αρχικά πολύ θετικές απέναντι στις ποσοστώσεις. Ε, βλέπουμε όμως ότι έχουν, αυξη... έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια, παρότι συνεχίζουν να αποτελούν μειονότητα στις θέσεις αυτές, 25 έως 40% σήμερα και έχουν περισσότερες θέσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις από ό,τι στις ιδιωτικές. Μόλις ε, το 6% των ε, διευθυντών εταιριών είναι γυναίκες. Και σας ε, ανέφερα πριν ότι η αγορά εργασίας είναι διαχωρισμένη ανάμεσα στα δύο φύλλα και μέχρι τώρα γυναίκες δεν εισέρχονταν σε ανδρικούς τομείς. Βλέπουμε όμως αλλαγές και ιδιαίτερα στη στάση των ανδρών απέναντι στις οικογένειές τους ε, και τα παιδιά. Ε, ιδιαίτερα από το 2000 που είχαμε την ε, νομοθεσία για ίση γονεϊκή άδεια για τους άντρες και τις γυναίκες, για, τους, για μητέρες και τους πατέρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαιτούνται αλλαγές και από την πλευρά των ανδρών και από την πλευρά των ε, ανδρών ε, για να πετύχουμε ισότητα. Το 90% των πατέρων ε, έχει αποφελθεί από τη δυνατότητα τρίμηνης γονεϊκής άδειας και βλέπουμε με, πιο ίση κατανομή της φροντίδας των παιδιών ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Στόχο τη νομοθεσία, λοιπόν, είναι ο πιο ίσω καταμερισμό τη δουλειά στο σπίτι καθώ και τη πιο ίσης θέσεις ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα των ανδρών, περνώ στην βία εις βάρος των γυναικών και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην επανάσταση μη του που συγκλώνησε την Ισλανδία. Μπορεί να ε, βρισκόμαστε σε ηγετική θέση τα τελευταία εννέα χρόνια όσον αφορά την ε, ισότητα των δύο φύλων. Ωστόσο, ο σχετικός δείκτης δεν ε, συμπεριλαμβάνει το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Η επανάσταση λοιπόν μη του ξεκίνησε ουσιαστικά στις 24 Νοεμβρίου 2017 όταν δημοσιεύτηκαν πάνω από 130 ιστορίες παρενόχλησης και βίας σε θέσεις εξουσίας και έκτοτε όλο και περισσότερες γυναίκες μίλησαν για τα περιστατικά που έχουν ζήσει όσον αφορά την παρενόχληση, την βία λόγω φίλου. Ήταν πολύ συγκλονιστικές κάποιες από τις ιστορίες αυτές. Και δύο, ιδιαίτερα, ε, ε, δύο ομάδες ιδιαίτερα με ε, συγκλώνησαν που είναι οι γυναίκες μετανάστες και οι γυναίκες στον αθλητισμό. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με νέο σχέδιο δράσης για την βελτίωση του χειρισμού τέτοιων ε, αδικημάτων. Θα υπάρξει σχέδιο ενίσχυσης ε, των ποινικών διαδικασιών ε, για βελτίωση της θέσης των θυμάτων και αναβάθμιση και συντονισμός των σχετικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Το νομικό περιβάλλον στο οποίο διεκπεραιώνονται τα σεξουαλικά αδικήματα θα επανεξεταστεί για βελτίωση της ε, θέσης ε, των ε, θυμάτων. Γνωρίζετε επίσης ότι θα επικυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα είμαστε το 30ο έτος που θα επικυρώσει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ε, είμαστε ναι, μάλλον η 30η χώρα που υπέγραψε τη σύμβαση, αλλά θέλουμε αρκετό καιρό για την ε, εφαρμογή της. Ο πρόεδρος της Ισλανδίας, Κοίνι Γιουχάνεσον, ε, μας στήριξε στην προσπάθεια αυτή. Είπε στην φετινή του πρωτοχρονιατική ομιλία ότι μπορεί να θυμόμαστε το 2017 λόγω του ότι οι γυναίκες ξεκίνησαν τον αγώνα κατά της βίας λόγω φύλου και ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτή η υποστήριξη για μας είναι θέμα κλειδί, διότι οι άντρες θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Οι γυναίκε ηγούνται του αγώνα για την ισότητα των δύο φίλων εδώ και δεκαετίες, αλλά σημαντικό είναι και οι άντρες να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές. Θα πρέπει να γίνουμε συνυπεύθυνοι, διότι οι γυναίκε ακόμα ασχολούνται με θέματα ισότητα των δύο φύλων, ενώ οι άντρε βρίσκονται σε περισσότερε ηγετικέ θέσει. Θέλουμε λοιπόν ε, αυτοί που χαράσουν πολιτική, αυτοί που λαμβάνουν αποφάσει, να συμμετέχουν με ε, πιο ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε την ε, πρωτοβουλία Barbershop, να συμμετέχουν δηλαδή οι άντρες περισσότερο. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι, το πρόβλημα, ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εδώ δεν είναι να αποκλείσουμε τις γυναίκες, είναι να πετύχουμε τη συμμετοχή και των ανδρών. Μπορεί να επικρίνει κανείς ε, το θέμα αυτό, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου και οι άντρες να μπορούν να συζητούν ε, το θέμα της ε, ισότητας των δύο φύλων. Η πρώτη διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το 2015 με πάνω από 500 συμμετέχοντες ε, και ήταν η πρώτη φορά που τόσοι άντρες υψηλού επίπεδου συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ για, για μια συζήτηση για την ισότητα των δύο φύλων. Με βάση τις επιτυχίες αυτής της εκδήλωσης και η Ισλανδία συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και στην έδρα του ΝΑΤΟ εδώ στις Βρυξέλλες και στη Γενέβη στον ΟΗΕ. Και θα ήθελα να αναφέρω, επειδή αναφέρθηκα ε, στην καμπάνια Me Too και τις γυναίκες στην πολιτική, μέχρι πρόσφατα το το 90% είχαν συμμετάσχει σε εκδήλωση Barbershop όπου απάντησαν στην ε, εκστρατεία μιτού και συζήτησαν ε, επί μια ολόκληρη μέρα πώς θα προσεγγίσουν το μιτού Το 90% λοιπόν των βουλευτών από όλα τα κόμματα, των ανδρών βουλευτών από όλα τα κόμματα συμμετείχε. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία και από τον ε, Δεκέμβριο ο πρόεδρος της ε, Ισλανδίας συμμετέχει στην ε, εκστρατεία του ΟΗΕ που λέγεται η φωσή και στόχο έχει να πετύχει τη συμμετοχή των ανδρών στις εκστρατείες ισότητας. Επίσης πριν δύο εβδομάδες έγινε επίσημος προτέκτορας του Ισλανδικού της Ισλανδικής Οργάνωσης ε, για ε, ομοφιλόφιλους ε, και ήθελα να το αναφέρω αυτό διότι θα πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα και αυτό έχει συμβάλει και στην πρόθεση των γυναικών, έχει, έχει οδηγήσει στην πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔ, λεσβιών, ομοφιλόφιλων κλπ. Ε, προσλέπω στη συζήτηση μετά από την ομιλία μου. Θα ήθελα όμως επίσης πολύ σύντομα να αναφερθώ στις σχέσεις ανάμεσα στην Ισλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Ε, γενικά ε, σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο στο θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντικό εταίρο κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών ε, στο διεθνές σκηνικό, για παράδειγμα στον ΟΗΕ. Πιο πρόσφατα Συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να ε, τονίσουμε το θέμα του παγκοσμίου εμπορίου και της ισότητας των δύο φύλων. Έχουμε φυσικά την ε, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που προβλέπει συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά και τις χώρες ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από την άλλη, την Ισλανδία, την Νορβηγία και το Λίχτενστάιν. Κάποιε νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των δύο φύλων έχουν συμπεριληφθεί στην συμφωνία. Τέλος, ε, θα ήθελα να αναφέρω ότι η ισότητα των δύο φύλων στηρίχθηκε και στηρίζεται μέσω του δημοσιονομικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που χρησιμοποιούν ε, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λίχτενστάιν για να μειώσει τις ε, οικονομικές διαφορές στην Ευρώπη και σε διμερείς σχέσεις. Και αυτό από μόνο του νομίζω ε, θα αποτελούσε ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση εδώ. Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν της Ισλανδίας ε, για την ισότητα των δύο φύλων είναι ότι δεν έρχεται από μόνη της, ε, απαιτεί σκληρή δουλειά, συλλογική προσπάθεια. Και αυτό οδηγεί σε πολιτική βούληση και την ανάπτυξη εργαλείων όπως είναι η νομοθεσία, ο προϋπολογισμός και η ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε διάφορες πολιτικές όπως είναι και το πρότυπο για την ίση αμοιβή. Παρά λοιπόν όλα αυτά, δεν είμαστε ο παράδεισος της ισότητας, παρόλα αυτά εργαζόμαστε με αυτόν τον στόχο και αυτή είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι πολύ ευχαρίστω θα ακούσω τις θέσεις της Επιτροπής σας και επίσης θα χαρώ να εξερευνήσουμε μαζί τρόπους συνεργασίας για να πετύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσω σουηδικά. Αν λοιπόν δεν καταλαβαίνετε σουηδικά, θα πρέπει να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ένα τον άλλον. Διότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές εμπειρίες στις εργασίες μας για την ισότητα. Και κατόπιν έχουμε και τις χώρες ΕΖΕΣ που επίσης ανήκουν στην οικογένειά μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να παρακολουθούμε τις εμπειρίες ο ένας του άλλου και να μην προσπαθήσουμε να επαναφεύρουμε τον τροχό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ισλανδία. Είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό, διότι ήμουν αντιπρόεδρος της αποστολής ΣΥΝΕΑ. Και πρόσφατα που βρέθηκα στην Ισλανδία, εξέτασα αυτήν την νέα νομοθεσία που στόχο έχει την ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Αυτό που σκέφτηκα εγώ πολύ, διότι ακούγεται σαν παραμύθι. Είχαμε συζήτηση σήμερα πόσο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ίσης αμοιβή. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις μισθολογικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση. Ήταν απλό το ταξίδι σας, ήταν εύκολο, είχατε πολλές συζητήσεις. υπήρχαν άνθρωποι αντίθετοι με την πρόταση αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια άλλα θέματα. Όπως είπα, είχαμε νωρίτερα τη συζήτηση σχετικά με το μισθολογικό χάσμα. Συχνά λέμε ότι πρέπει να φροντίσουμε οι γυναίκες να εισέλθουν στα ανδρικά επαγγέλματα. Θα πρέπει οι γυναίκες τότε να εκπαιδευτούν για να εργάζονται στις δουλειές αυτές και να βγάζουν πολλά λεφτά. Ενώ δεν δεν λέμε ότι πρέπει να αυξήσουμε το μισθό σε τομείς γυναικείους, διότι θέλουμε και άντρες στην φροντίδα ε, των παιδιών, στον τομέα της υγείας ε, κλπ. Είχατε και τέτοιες συζητήσεις στην Ισλανδία. Και τέλος, το τελευταίο που είπες σχετικά με τους άντρες στην Ισλανδία. Είπες ότι οι άντρες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για ισότητα βλέπουμε στην επιτροπή μας ε, που συζητάει με τα θέματα αυτά πολύ συχνά ε, νιώθουμε πολύ μόνες, μόνο γυναίκες έχουμε εδώ και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι και οι άντρες να συμμετέχουν στις εργασίες αυτές, διότι στο κοινοβούλιο έχουμε περισσότερους άντρες από ό,τι γυναίκες. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί οι άντρες στην Ολομέλεια δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις, για μια Ευρώπη ίση δεν θα πετύχουμε την ισότητα. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το ότι και οι άντρε τη Ισλανδία έλαβαν την απόφαση αυτή και ελπίζω να μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο και εδώ στην Ευρώπη. Αυτέ λοιπόν ήταν οι ερωτήσει μου και δίνω τώρα το λόγο σε, σε άλλες ευρωβουλευτίνες αν έχουν ερωτήσεις προς την πρέσβη της Ισλανδίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου, Άννα. Πού είναι οι άντρες? Πάντως στην Επιτροπή μας λάμβονται τις απουσίες τους. Πού είναι οι άντρε όταν συζητούμε τόσο σημαντικά πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα-δύο το πολύ παίρνουν το λόγο, παρά το μεγάλο αριθμό του στην Ευρωβουλή. Κυρία Πρέσβυρα, ποιο είναι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού τη Ισλανδία. Επίσης, για το εκπαιδευτικό σας σύστημα. Η παιδεία σας ήδη από την παιδεία δίνει έμφαση στην ισότητα των φύλων, ήδη από την παιδική ηλικία. Επίσης, ε, η πολιτική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ε, κρατικές πολιτικές. Επίσης, τι επίπεδα έμφυλης βίας έχετε στην Ισλανδία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε και τέτοια στοιχεία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Πρέσβη για την παρουσίασή της. Θα ήθελα επίσης να τη συγχαρώ για τα όσα έχετε πετύχει στο θέμα αυτό στην Ισλανδία. Στο θέμα δηλαδή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να τονίσω έναν τομέα, τη συμμετοχή στην πολιτική. Είναι απίστευτο το ότι έχετε πετύχει η ισότητα αν και είπατε ότι ανάλογα με τις εκλογές υπάρχουν διακυμάνσεις αλλά είχατε φτάσει σχεδόν το 50% όσον αφορά τη συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Πολλές θεωρητικές συζητήσεις γίνονται σε δημοσιογραφικό επίπεδο, αλλά και σε άτυπες συζητήσεις. Πώς επηρεάζει αυτό τις πολιτικές αποφάσεις μιας χώρας όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό γυναικών στην λήψη αποφάσεων. Είστε διπλωμάτης, έχετε βρεθεί σε πολλές χώρες όπου δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, όπου δεν εκπροσωπούνται τόσο καλά οι γυναίκες στην πολιτική. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις εμπειρίες σας. Πώς διαμορφώνεται διαφορετικά η πολιτική όταν πετυχαίνετε η αναλογία 50-50% στο Κοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Επομένως, σας δίνω και πάλι το λόγο. Κύριε Πρέσβη, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να απαντήσω εύκολα σε όλα. Θα βάλω τα δυνατά μου. Πάντως, θα ξεκινήσω με τις δικές σας ερωτήσεις πρώτα, λέει στην Πρόεδρο. Σε ό,τι αφορά τις ίσες αμοιβέ, το πρότυπο για τις ίσες αμοιβέ. δεν υπήρχαν μεγάλες συζητήσεις και διαφωνίες σε ό,τι αφορά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο. Οι, οι διαφωνίες είχαν να κάνουν με το κατά πόσο έπρεπε να είναι νομοθετημένο. Με συνεργασία όμως μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και των διαφόρων συνδικάτων αλλά και της κυβέρνησης, όλοι αυτοί οι φορείς εργάστηκαν από κοινού για να αναπτύξουν αυτό το πρότυπο, αλλά όταν έφτασε η ώρα να θεσμοθετηθεί νομικά, αυτό ήταν το μόνο αρνητικό σημείο, θα έλεγα, όλες αυτές οι διαφωνίες. Όχι όμως το να υπάρχει ένα πρότυπο. Σε γενικές γραμμές πιστεύω όμως τώρα ότι υπάρχει ικανοποίηση από όλες τις πλευρές και από τους περισσότερους βουλευτές, οι οποίοι συμφωνούν για την υποχρεωτική φύση του προτύπου αυτού του μισθολογικού. Αλλά όπως σας είπα υπήρξαν κάποιες φωνές εναντίον αυτής της υποχρεωτικής φύσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή των ανδρών περισσότερο στην οικογένεια και στην ανατροφή των παιδιών αλλά και στη φροντίδα των παιδιών γενικά, το ζήτημα αυτό προέκυψε με την γονική άδεια που έκανε τεράστια διαφορά διότι δεν υπήρχε μονάχα η αδιαμητρότας, η μητέρα που θα έπρεπε να φροντίσει τα πολύ νέα παιδιά, αλλά και ο πατέρας. Όπως είπα, αυτό τελικώς απεδείχθη μια πολύ θετική α, ένα πολύ θετικό βήμα με εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις. Το γεγονός δηλαδή ότι και οι πατέρες μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την άδειά τους όταν γεννήθηκαν τα παιδιά τους. 90% των ανδρών, όπως είπα, χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα αυτή της γονεϊκής άδειας. Μιλήσατε και για τον διαχωρισμό στον εργασιακό χώρο και πώς υποτιμούμε και δεν δίνουμε σημασία στις παραδοσιακά γυναικείες εργασίες. Στόχος μας είναι να επανεκτιμήσουμε το πώς εξετάζουμε τι διάφορε δουλειέ. Ποιε δουλειέ θεωρούνται σημαντικέ, ποιε δουλειέ θεωρούνται λιγότερο σημαντικέ. Επομένω, μακροπρόθεσμα, στόχο μα θα ήταν και αυτό, η επανεκτίμηση των γυναικείων εργασιών. Αυτό όμω είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Στην Ισλανδία, για παράδειγμα, δύο τρίτα των σπουδαστών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκε. αλλά αυτό δεν αντανακλάται στου μισθού αναγκαστικά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μακροπρόθεσμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φτιάξουμε. Η εκτίμηση, αξιολόγηση των εργασιών είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση από μόνη της. Στην Ισλανδία υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα που απεργούν γιατί θεωρούν ότι δεν χαίρουν εκτίμησης σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Βλέπουν τα πολύ υψηλό, υψηλό στελέχη να έχουν υπέρογους μισθούς Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τομέας ε, εν στον οποίο πρέπει να εργαστούμε. Ρωτήσατε και για το πρόγραμμα Barbershop. Όχι, δεν υπήρχε ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική, σας είπα ότι είναι μια μάχη που μένετε στις εκλογές όπου ο αριθμός των γυναικών από 48% έφτασε στο 38% είναι, δεν είναι ακόμα σταθερό το πολιτικό επίπεδο και ακόμα αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις οικονομικής κρίσης του 2008. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε αρκετά μικρά νέα πολιτικά κόμματα Και επίσης έχουμε και κόμματα των άκρων. Και έχουμε και μικρότερη συμμετοχή γυναικών σε αυτού του τύπου τα κόμματα, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη σύσταση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει και πάλι να βρούμε την ισορροπία μας και ε, να αυξηθεί και πάλι η συμμετοχή των γυναικών. Σας είπα ότι φτάσαμε σχεδόν το στόχο του 50%. αναφορικά με τη διαφορά των συνθήκων στις διαφορετικές χώρες. Κάθε χώρα έχει τις δικές της παραδόσεις, κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία. Και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μιας χώρας σε μια άλλη χώρα έτσι απλά. Είναι ανάγκη να προσαρμοζόμαστε. Αυτό που είναι σημαντικό Μπορεί κανείς να πει ότι τα θέματα των δύο φύλων είναι κάτι το οποίο πλέον έχει εισχωρήσει στην πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Η συζήτηση έχει να κάνει με το πώς θα φτάσουμε εκεί. Κάποιες χώρες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση ίσως το περιορισμένο μέγεθος της χώρας μας να λειτουργήσε προς οφελό μας, γιατί η κοινωνία λειτουργούσε με πιο διάφανο τρόπο σε γενικές γραμμές, ήταν πιο εύκολο να δούμε τι συμβαίνει. Πιστεύω είναι δύσκολο να πούμε με ποιον ακριβώς τρόπο οι άλλες χώρες θα πρέπει να δράσουν. Ίσως να υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα και για άλλες χώρες. έχω σε ό,τι αφορά την ισότητα που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία και τις πολιτικές που αφορούν τα φύλλα να είναι παρούσες σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές, όλες οι πολιτικές της κυβέρνησης, όλες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτό το στοιχείο τις, να τις εξετάζουμε υπό το, υπό το πρίσμα της ισότητας των δύο φύλων. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι όλες οι, οι πολιτικές προσαρμόζονται σε αυτό το, το ζητούμενο της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Αναφορικά με την σχολική διδασκαλία, αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, αναπτύσσεται ένα τέτοιο πρόγραμμα. η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων θα είναι ένα σημαντικό μάθημα που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Και με αυτά πιστεύω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις σας, λέει η πρέσβης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε την εμπειρία σας στην Ισλανδία και το έργο που κάνει η χώρα αυτή υπέρ της ισότητας των φύλων. Ελπίζω την επόμενη διετία να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το, το βαθμό εφαρμογής ε, της σχετικής νομοθεσίας. Και ελπίζω να μιμηθούμε το παράδειγμά σας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ισότητας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Και να προσθέσω ότι αν υπάρχουν ειδικά θέματα που σας ενδιαφέρουν, γιατί εγώ ακροθυγός μίλησα για πολλά, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν πρόλαβα να καλύψω. Αν έχετε απορίες, είμαστε στη διάθεσή σας και θα έρθουμε με την ίδια ευχαρίστηση και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Okay, we have some more work to do before... Έχουμε και άλλα θέματα. Πριν διεκπαιρεώσουμε την απογευματινή μας συνεδρία, είμαστε στο σημείο 6, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1303 του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και αλίες και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας και για την κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Σύρπα Πιετικά, είναι από το ΕΛΚ, στην οποία δίνω και το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ήταν τόσο εντυπωσιακό και μακροσκελή ο τίτλο ε, και εισαγωγή που κάνατε για την έκθεση. Σα ευχαριστώ. Το περιεχόμενο είναι ε, πιο συνοπτικό από τον ίδιο τον τίτλο. Πάντω η ουσία είναι σημαντική. Γιατί τα... Βέβαια τα χρήματα είναι χρήματα και χωρίς τη διάσταση του φύλου ε, και τα διά, οι υποδομές είναι το ίδιο και η υγεία είναι το ίδιο και όμως δεν ισχύει αυτό. Γιατί σίγουρα ο οικονομικός και δημοσιονομικός ε, παράγοντας είναι ουδέτερος από άποψη φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι είδους κοινωνίες διαμορφώνουμε και τι ε, πολιτική φύλου προωθούμε με τις ε, δημοσιονομικές και οικονομικές μας πολιτικές. Γι' αυτό προτείνουμε ε, μια μεγαλύτερη διαφάνεια για να είναι προφανές τι στηρίζουμε. Και γι' αυτό κρίνω σημαντικό να γίνει μια ανάλυση και μια αξιολόγηση του αντικτύπου του φύλου. Και πριν να γίνει οποιαδήποτε δημοσιονομική οικονομική πρόταση να προηγείται μια μελέτη ε, αντικτύπου φύλου. Για μερικούς είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι θα πρέπει να δούμε. Οι γυναίκε είναι οι άνδρες που χρησιμοποιούν περισσότερο τα γιοταχή του. Αυτό το θέμα θα επηρεάσει την απόφαση για τις επενδύσεις οδικέ μεταφορές. Ε, πως οι γυναίκε χρησιμοποιούν περισσότερο τις αστικές συγκοινωνίες ή τους σιδηροδρόμους. Άρα θα υποφεληθούν καλύτερα από βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ή τη αύξηση των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων οι άνδρες ή οι γυναίκες εποφελούνται περισσότερο ή ε, έρχονται σε δυσμενή θέση λόγω της χειρότερης λειτουργίας του συστήματος παροχής ε, φροντίδος στην τρίτη ηλικία. Ποιος εποφελείται περισσότερο ε, για τη συνδυασμό του επαγγελματικού με το προσωπικό του βίο. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μία ανάλυση από τη σκοπιά του φίλου πάντα πριν την χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής. Αυτό που είναι σημαντικό και το έχουμε επανειλημμένω δηλώσει στην Επιτροπή είναι η ιδέα του προπολογισμού από τη σκοπιά του φύλου. Όχι μόνο σε επίπεδο ανάλυσης, αλλά θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδου δημοσιονομικέ αρχές όπου θα προωθούμε αυτή την έμφυλη διάσταση και να δούμε ποιο φύλλο αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα ή που εκπροσωπείται ή δεν έχει αποφεληθεί ή δεν έχει ευνοηθεί από συγκεκριμένα κονδύλια του προϋπολογισμού. Κάτι που χαιρετίζουμε ήδη στα ταμεία είναι η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς για την ισότητα των φύλων. Έχουμε μια κατάρτιση σχετική υπέρ της ισότητας των φύλων για το προσωπικό και τα ηγετικά στελέχη της ΕΙΕΔ ε, και το θεωρούμε προϋπόθεση για την έγκριση, ισότητα των φύλων, προϋπόθεση για την έγκριση εθνικών προγραμμάτων. Θα πρέπει όμως και το προσωπικό να είναι καταρτισμένο ανάλογα πριν προσαρμοστούν τα κονδύλια και τα προγράμματα στην εθνική πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια πολύ σημαντική προϋπόθεση που ελπίζω να επεκταθεί ε, σε όλα μας τα ταμεία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της έκθεσης μου. Δεύτερο. Η Επιτροπή και τα κρατημέλη θα πρέπει να μερεμνήσουν ώστε η πρόταση να μην οδηγεί σε περικοπή των διαθέσιμων πόρων και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα των Φύλων ή τη στρατηγική δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων και θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα προγράμματα για τα ταμεία να έχουμε ορόσημα για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν την ισότητα των φύλων. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει να διδαχθούμε από ε, τη Τη μέχρι τώρα εμπειρία μα και τα υφιστάμενα προγράμματα, γιατί δεν είναι μακροσκελή ο κατάλογος των ταμείων. Να δούμε τι προγράμματα και τι σχέδια στηρίξαμε μέχρι τώρα. Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες μελέτες που δείχνουν ότι προτεραιότητες όπως η παροχή φροντίδας, οι προσβάσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, οι αστικές συγκοινωνίες, η πρόσβαση στην Ήπεθρο και όλα αυτά δεν έχουν αναγνωριστεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί. Αυτό θα πρέπει να είναι ο, αυτός θα πρέπει να είναι ο γνώμονάς μας, κυρία Πρόεδρε. Αυτό θα πρέπει να διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αυτό να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Να τηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις και τα κονδύλια όλα αυτά να εξυπηρετούν και το στόχο της ισότητας των φύλων. Και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα ταμεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πιέτε Κάινεν. Δεν θέλει κανείς το... Δεν βλέπω κανένα από τους πιο δυσηγητές μάλλον. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο για το σημείο αυτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχής είναι ο το μόνο εργαλείο, ο μόνος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την ε, πρόθεση της κοινωνική και ταφικής συνοχής. Και η αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να έχει στόχο τη βελτίωση και όχι την επιδείνωση ή ε, στασιμότητα της πολιτικής συνοχής. Και η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να ζητήσει ε, μέτρα σαν αυτά που υιοθέτησε η Ισλανδία να γενικευθούν για να ε, λαμβάνεται υπόψη η πολιτική των φύλων και στην πολιτική συνοχή και σε άλλες πολιτικές. Να είναι αναπόσπαστο στοιχείο όλων των πολιτικών. Επίσης, συμφωνούμε με την μελέτη επιπτώσεων των πολιτικών ε, ε ως προς την έμφυλη τους διάσταση πριν γίνει η κατανομή των κονδύλιων και οι διαχειριστές των κονδύλιων θα πρέπει να μεριμνούν για το γεφύρωμα του μισθολογικού χάσματος, για την ισότητα των φύλων, για την προστασία των ανέργων γυναικών, των συνταξιούχων ή την προστασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, που δημιουργούν γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ευαισθησία για όλα αυτά τα θέματα και να μην ε, ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ισότητα των φύλων είναι εθνική αρμοδιότητα και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και του ευρωπαϊκού μηχανισμού, όπω την πολιτική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνθήκων θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα θέματα, αλλά και τα κρατημέλη οφείλουν να εφαρμόζουν την αρχή τη ισότητα των φύλων και τη πάταξη των διακρίσεων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε μαχητικοί και στο θέμα της μακροαιρεσιμότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα μέτρα λιτότητας έπληξαν πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του κανονισμού και υπέρ της ε, εισαγωγής θετικών στοιχείων στο κείμενο, αλλά όχι πάση θυσία βέβαια, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δω αν είναι κανείς παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να θέλει να πει κάτι. Όχι. Να ξαναδώσω το λόγο στη ΣΥΡΠΑ, αν θέλει να ξαναπεί κάτι, αν θέλει να ξαναπάρει το λόγο. I just would like to... Θα ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας. και να ευχαριστήσω την Γραμματεία και τους άλλους ευρωβουλευτές για τη συμβολή τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 13 ε, ε, Ιουλίου 2018 φέτος, 12 η ώρα το μεσημέρι και κατόπιν έχουμε ψηφοφορία εδώ στην ΦΑΜ στις 3 Σεπτεμβρίου και την ψηφοφορία στην Επιτροπή Ρέγγι στις 9 Οκτωβρίου. Προχωράμε τώρα στην τελευταία έκθεση για σήμερα σχετικά με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Γιώργη Σολέ είναι η συγγήτρια από τους Πράσινους. Thank you, Madam Chair. Ο Γιώργη Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαρίστω σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση για την πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Μια γενική παρατήρηση. Στηρίζω απόλυτα την δημιουργία αυτής της αρχής που θα βελτιώσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εργασιακού και Κοινωνικού Δικαίου. Θα προωθήσει την διασυνορική κινητικότητα θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού κοινωνικού, της διασυνοριακής κοινωνικής ε, απάτης και θα βοηθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων. Όσον αφορά την ε, τυχή της ισότητας των δύο φύλων στη γνωμοδότηση αυτή, οι γυναίκες συγκεντρώνονται δυσανάλογα και συχνά μη ηθελημένα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα που να εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και σε αυτόν τον τομέα. Ε, και στο πλαίσιο αυτής της νέας αρχής. Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, και κατά την εφαρμογή του κύκλου πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, προτείνω να ε, ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου με τη χρήση δικτών ε, και κατά την, ε, τον ετήσιο και τον πολιετή προγραμματισμό της αρχής αυτής. Επίσης, ε, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου, καθώς και κατά την συλλογή δεδομένων. Να συμπεριληφθούν ξεχωριστά κεφάλαια για την ισότητα των δύο φύλων στις ετήσιες εκθέσεις και ε, στην παροχή πληροφοριών ε, σε ε, άτομα και σε επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας σχετικά με, για παράδειγμα, τις γονεϊκές άδειες. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει ανάλυση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την ισότητα των φύλων να συμπεριλαμβάνονται επίσης οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στην ομάδα των συμφεροντούχων και να διασφαλίζεται η ισορροπημένη από πλευράς φύλου σύνθεση της αρχής αυτής, καθώς και στους συμβουλευτικούς φορείς. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις, ε, αυτές είναι οι ιδέες που θέλω να παρουσιάσω στην ομοδότηση αυτή και πολύ ευχαριστώ θα ακούσω τις ε, παρατηρήσεις σας και τους προβληματισμούς σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Δεν έχουμε κανέναν από το ΕΛΚ. Έχουμε όμως τη Μαρία Αρένα που θα μιλήσει στο όνομα της ε, Δίλια Πλινκεβιτσιούτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, παίρνω το λόγο για τη σκιώδη εισηγήτρια, την οποία και αντικαθιστώ σήμερα η Μπίλια συμφωνεί με όσα Υπόθεκαν σε ό,τι αφορά τον ρόλο της αρχής, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την εργασία. Μπορούμε να, χαρούμε για μια τέτοιου τύπου αρχή. Εξ αρχής όμως πρέπει να θέσουμε το ζήτημα της νομότητας μεταξύ ανδρών και γενικών στη δημιουργία αυτής της αρχής. Θα είναι δύσκολο να επανέρθουμε, επομένως πρέπει να χτίσουμε εξ αρχής σωστά είναι ανάγκη σε ό,τι αφορά την διαχείριση της αρχής αυτής να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην εγκατάσταση της αρχής αυτής. Το δεύτερο έχει να κάνει με την διάσταση της αρχής αυτής. Θα εργάζεται εναντίον των καταχρήσεων, θα θα πρέπει επίσης να ενημερώνει τα άτομα για τα δικαιώματά τους. Έχουμε σε τεράστιο βαθμό γυναίκες, μιλάμε συχνά για κινητικότητα μεταξύ των ανδρών εργαζομένων, όχι όμως για τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά το τομέα της φροντίδας ή της συνοδείας ατόμων, υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες οι οποίες μπορούν να, να κινηθούν, αλλά δουλεύουν σε συνθήκες σε ό,τι αφορά τα συμβόλα εργασίας τους, σε ό,τι αφορά την ε, βεβαιότητα. Αναφέρομαι στις ε, γυναίκες ε, που, εργαζόμενες που κινούνται στο εσωτερικό της Ευρώπης. Είναι ανάγκη λοιπόν να τις ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, να βελτιώνουμε την κατάσταση της χώρας από την οποία προέρχεται η κάθε τέτοιου τύπου εργαζόμενοι. Είναι ανάγκη να προσφέρουμε βοήθεια και ε, στους κοινωνικούς εταίρους, στα συνδικάτα. Η Μπιλιά λοιπόν χαίρεται ιδιαίτερα που εργάζεται από κοινού μαζί με τον εισηγητή για να μπορέσει να προτείνει και ε, τροπολογίες επικοδομητικές ε, έχοντας στο μυαλό τις ανάγκες των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Μαρία. Και τώρα η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και από μένα να σταματήσω να μιλάω συνέχεια. Σε ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Σόλη στις προτάσεις που το είδαμε μέσα από το προσχέδιο της γνωμοδότησης που συνέταξε. Βρίσκεται σε μια καλή κατεύθυνση. Κανείς δεν τα εμφιβάλλει αυτό. Όμως δεν αρχεί η ένταξη δικτών με βάση το φύλλο, όπως προτείνει ο εισηγητής, ούτε η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας στη διαδικασία δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας θα βοήθησε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και μην πει κανένα ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασία και άρα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Στην Ευρώπη, το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασία αυξήθηκε στο 50,9% σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις τάσεις στην αγορά εργασία για το 2017. Το ποσοστό αυτό είναι 13 μονάδες, 13 μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο του αντρικού εργατικού δυναμικού. Αν μέχρι το 2025 καταφέρναμε να κλείσουμε την ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασία, θα προσθέταμε περίπου 410 δισεκατομμύρια στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, γιατί στερείται αυτό το γενικό εργατικό δυναμικό να μπει στην αγορά εργασία, γιατί στερείται το δικαίωμα στην εργασία, να σας προλάβω. Δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασία, δεν είναι γιατί είναι επιλεκτικές ω προ τις θέσεις εργασία, ούτε του λείπουν δεξιότητε και προσόντα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Στερούνται μια αγορά εργασίας που στο επίκεντρο θα έχει την ισοτιμία, τη σταθερότητα, την, αξιο, την αξιοκράτεια, την αξιοπρεπία και την προστασία που χρειάζονται οι εργαζόμενοι ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να τους εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Όταν ανακοινώθηκε επίσημα η πρόταση της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, ο Επίτροπος Τίμερμαν ανέφερε συγκεκριμένα το έργο μας για την διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού ολοκληρώνεται με την σημερινή πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αυτό είναι σημαντικό για την σωστή λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε κίνηση για την εξέβρεση των κατάλληλων πληροφοριών και θα ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την επιβολή δικαίων και αποτελεσματικών κανόνων, μας είπε ο Τίμερμανς. Βλέπετε στην παραπάνω δήλωση να αναφέρεται κάπου η προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε να λέει πως θα διασφαλίζει η αρχή δίκαιες συνθήκες εργασίας για τα μετακινούμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργατικό δυναμικό. Βλέπετε να προάγει την ισότητα και την ισοτιμία μεταξύ εργαζομένων. Ανάμεσα στους 17 εκατομμύρια πολίτες που μετακινούνται για εργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζεται μια ισοδυναμία αντρών και γυναικών 50-50. Αυτό είναι εκ πρώτης όψιος καλό. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στις λεπτομέρειες, θα δούμε τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στις χώρες προέλευσης των μετακινούμενων. Για παράδειγμα, ενώ πάνω από 60% των μεταναστών μετακινούμενων από τη χώρα μου, την Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία, είναι γυναίκες. Στη Ρωμανία και την Πολωνία αυτό το ποσοστό είναι κάτω από 25%. Πού οφείλεται αυτές οι τεράστιες διαφορές και τι επιπτώσεις έχουν στα ιδιαίτερα δικαιώματα προστασίας των εργαζομένων γυναικών. Αντίστοιχες τεράστιες διαφορές υπάρχουν και στις εισρωές μετακινούμενων εργαζομένων αναχώρα. Στην Ελλάδα είναι γυναίκες το 55% των μετακινούμενων εργαζομένων από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν στη Λιτουανία το ποσοστό τους είναι μόλις 25%. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το παράδοξο. Μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Το μυστικό είναι οι εξασφαλισμένα χαμηλότερες αμοιβέ των γυναικών. Για παράδειγμα, στη Γερμανία θα πάνε νοσοκόμες ή φροντίστριες ασθενών από την Ελλάδα, πρόθυμες να πληρωτούν λιγότερα. Στην Ελλάδα θα έρθουν εργαζόμενες από τη Βουλγαρία ή τη Ρωμανία που θα δουλέψουν στο τουριστικό κλάδο με ελάχιστες αμοιβέ και χωρίς δικαιώματα ακόμα και τελείως αντίλωτες. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χρειαζόμαστε μια διακοσμητική Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που απλώς θα καταγράφει τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο. Χρειαζόμαστε μια υποπτική αρχή που θα διασφαλίσει πως το υπάρχουν κοινοτικό δίκαιο τα εφαρμόζεται. Αρχίζοντα, αρχίζοντας από την οδηγία για την ίση αμοιβή, για ίδια εργασία από την καταγραφή και πάταξη της αντίλωτης εργασίας και των επισφαλών συνθηκών εργασίας, τα πρώτα θέματα των οποίων είναι οι γυναίκες. Χρειαζόμαστε μια αρχή που τα λαμβάνει στην εξάλληψη της διάκρισης με βάση το φύλλο, μια αρχή που θα προστατεύει τις έγκυος εργαζόμενους από απόλυση και τα επιβάλλει πρόστιμα στους εργοδότες και όχι το ανάποδο, χρειαζόμαστε μια αρχή που θα διασφαλίζει την τήρηση των ωραρίων και των συνθήκων ασφάλειας και υγιεινής στη δουλειά. Χρειαζόμαστε μια αρχή που στο επίκεντρο θα έχει το εργατικό δυναμικό και όχι το καπιταλιστικό αφεντικό. Να μην κάνουμε άλλη μια τρύπα στο κοινωνικό κενό που όλο και μεγαλώνει στην Ένωση. Να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να εφαρμόζουμε κανόνες για μια καλύτερη, δικαιότερη, εσφαλίστερη εργατική ζωή στην Ευρώπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Thank you, Σας ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Άλλος κανείς παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ουγγαρία δεν έχουμε πολύ καλές εμπειρίες από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάρος ε, ενός κράτους μέλους. Βλέπουμε ε, διακρίσεις. Όσον αφορά όμως ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, ε, σκέφτομαι ως νομικός και γι' αυτό ελπίζω, διότι μιλάμε για συγκεκριμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει η αρχή να ελέγχει την εφαρμογή αυτών των προτύπων. Αυτά τα εργασιακά πρότυπα βλέπουμε να παραβιάζονται και ιδιαίτερα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου εργοδότες ε, και, και από τις χώρες αυτές, αλλά και από την Δυτική Ευρώπη, εκμεταλλεύονται στιγνά την κατάσταση και την ισχύ τους. Εκμεταλλεύονται το εργασιακό δίκαιο και κάνουν πράγματα που ποτέ δεν θα μπορούσαν να κάνουν στις δικές τους χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνο με την προραλή σας και θα ήθελα να παριθμίσω κάποιες πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου θα πρέπει να γίνουν ενισχυμένοι έλεγχοι και να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Για παράδειγμα, υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο για τις υπεργολαβίες, αλλά πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή και αντί να συνάψουν συμβάσεις εργασίας μεγάλης διάρκειας εκμεταλλεύονται τους κανόνες. Αυτό ισχύει και για την ε, άσκηση των ε, εργαζομένων ε, πριν λήξει η, η περίοδος ε, άσκησης ε, τους απολύουν και προσλαμβάνουν καινούριου ασκούμενους. Βλέπουμε αυθαίρετες απολύσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν τηρούνται λοιπόν οι προϋποθέσεις εργασίας. και συχνά βλέπουμε διαφορετική κατάσταση υπό τον ίδιο δυτικο δυτικό-ευρωπαίο εργοδότη. Μια τέτοια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης και σε θετικές αλλαγές για τους εργαζομένους ε, στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Επιτροπή μας μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών. και οι γυναίκες που υφίστανται ακριβώς ε, τις χειρότερες διακρίσεις ε, μπορούν να δούνε καλύτερες ε, συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να θέλει να πάρει το λόγο, να δώσω το λόγο στον συντάκτη της νομοδότης, τον κύριο Ζόρντι. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τις τρεις συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και μας παρουσίασαν τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες τους. Και εγώ συμμερίζομαι ε, την ανησυχία σας ε, ως προς τη διαφορά στις εργασιακές συνθήκες ή σε μια αποκατάσταση μιας μεγαλύτερης δικαιοσύνης ε, στις εργασιακές συνθήκες μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Και στη δική μου χώρα θα ήθελα να έχουμε ισότιμες εργασιακές συνθήκες για όλους και ειδικώ για τις γυναίκες. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η γνωμοδότηση αυτή αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα επικεντρωθεί στην ε, διασυνοριακή κινητικότητα, στα διασυνοριακά ζητήματα. Και οι εύλογε ανησυχίε σα ε, τι οποίες και εστερνίζομαι, αφορούν περισσότερο την οδηγία για τις εργασιακέ συνθήκες την οποία προωθούμε στην ε, δική μου πολιτική ομάδα γιατί θέλουμε ε, ε, σαφή ελάχιστα πρότυπα και εργασίκες προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν πολλά κενά, πολλές αδυναμίες, ε, πολύ ατελής εφαρμογή των διατάξεων αυτών και χρειάζονται πιο αντατική έλεγχη. Πάντω στη γνωμοδότησή μου αυτή προσπαθώ να αποκαταστήσω μια ισορροπία μεταξύ των φύλων, μια συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και μια ισότητα των φύλων μέσω αυτής της ειδική αρχής, ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, που θα έχει εντολή που θα περιορίζεται ή θα εστοχεύει κυρίως στη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Ευχαριστώ πάντως για τις ε, παρατηρήσεις και προσβλέπω σε πολύ εργαστή συνεργασία στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, το χρονοδιάγραμμα τώρα. Ε, η διορία για την ε, υποβολή προ... τροπολογία ολίγη 12 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στις 27 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Γυναικών και στην Αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης, στις 18 Οκτωβρίου. Οπότε ολοκληρώσαμε την ε, απογευματινή ημέρη σε διάταξη. ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ κυρίως τους διερμηνείς. Καλό βράδυ σε όλους.